Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε στις θέσεις σα παρακαλώ, Κυρίε και κύριοι. αγαπητοί πρόεδρε τη ΑΕΜΑ, ε, του Κοινοβουλίου της Λετωνίας, κύριε Επίτροπε Μοσκοβισή, Οι συνάδελφοι Μόλτοβα και Αρτουή πιστεύω θα έρθουν σύντομα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην δεύτερη σύνοδο της διάσκεψης. Α, καλώς ήταν, κύριε μου. I welcome uh, Mr. the Vice President of the European Investment. ορίζω τον κύριο Μόλτερ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τον συνάδελφο πρόεδρο της Επιτροπής ε, ε, τον κύριο Αρτσουή. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε την κατάσταση σε σχέση με το Fiscal Compact και την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομικής Ένωσης. Αγαπητοί συναδελφοί από τα Εθνικά Κοινοβούλια, θέλουμε να ακούσουμε ποια είναι η δική σας εμπειρία στην εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, του Fiscal Compact. Θα θέλαμε να ακούσουμε εσείς τι άποψη έχετε. Ξέρετε ότι έγινε μια προσπάθεια για μια Δημοσιονομική Ένωση πέραν τον, ε, του ελέγχου του βουλευτού, των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Αγωνιστήκαμε για τα θέματα αυτά για να μείνουμε μέσα στην ε, διακοινωτική μέθοδο, στην κοινοτική μέθοδο, γιατί πιστεύουμε ότι η κοινοτική μέθοδος είναι και πιο δημοκρατική και πιο αποτελεσματική και αποτελεί την ε, συνταγή επιτυχίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εξισορροπεί τόσο το συμφέρον, τα συμφέροντα των μικρότερων με τα μεγαλύτερα κράτη, και εκείνων που έχουν περισσότερη ή μεγαλύτερη ή λιγότερη ευημερία ή των κρατών του Βορρά και του Νότου μπορεί να επιλύσει μέσω του διαλόγου και της συνένεσης τις διαφορές και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι κύριες διαδικασίες για τη δημοσιονομική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζονται στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Θετικό αυτό για πολλές δεκαετίες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητοί συναλφοί, ήταν η υπόσχεση της ειρήνης, της ευημερία. Και θέλουμε να ξαναγίνει αυτή η υπόσχεση η Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Απλώς θα πρέπει να προσέξουμε εξίσου με τα λοιπά θέματα την απασχόληση και τους κοινού δείκτες. Εξίσου δηλαδή με, τα, με τους δημοσιονομικούς και μακροοικονομικούς δείκτες. Πρόκειται για θέματα που αφορούν τον απλό άνθρωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρωνόταν στην εμβάθυνση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών πολιτικών μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής και νομισματικής ένωσης, αλλά ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την τήρηση των κοινωνικών δικτών, όχι μόνο των δημοσιονομικών κανόνων και πρέπει εξίσου να τιμωρείται η παραβίασή τους. Άρα λοιπόν ένας πίνακας αποτελεσμάτων όπως τον προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα για τους κύριους δείκτες της απασχόλησης και των, της κοινωνικής προστασίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην ε, εξισορρόπηση του πίνακα αποτελεσμάτων για τα δημοσιονομικά. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε για μια πιο ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Ήρθε η ώρα, πιστεύουμε, να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προστατεύει τον πολίτη τη μέσα από μια κοινωνική διάσταση, κυρίως καθώ ο πολιτή είναι Εκείνο, ο οποίο εξακολουθεί να πληρώνει το τίμημα τη οικονομική κρίση. Η Ευρώπη έχει, έχει περιπέσει σε έναν φαύλο κύκλο με χαμηλή ανάπτυξη, με ε, χαμηλά εισοδήματα που τροφοδοτούν την ανεργία και πως εκ τούτου τροφοδοτεί την ύφεση. Έχουμε ακόμα 35 εκατομμύρια ανέργους Ευρωπαίους, εκατομμύρια κινδυνεύουν από τη φτώχεια και κινδυνεύουμε πάνω απ' όλα όλοι να μείνουμε πίσω σε σχέση με τις ανταγωνιστικές χώρες εάν δεν κάνουμε κάτι αμέσως. Εμείς χρόνια τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούμε να υπάρξουν επενδύσεις που θα συμπληρώνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Ο πρόεδρος Γιουνκέρ ε, στις 26 Νοεμβρίου ε, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επενδύσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζουμε ολόκαρδα. Επενδύσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι είμαστε προσιλωμένοι σε μια Ευρώπη νέα με ανάπτυξη και με θέσει εργασίας. Καλούμεθα όλοι τώρα να αναλάβουμε τις ευθύνε μας και να εξασφαλίσουμε το δημοσιονομικό αυτό σχέδιο να έχει τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίε επιτυχίας. Αυτό πιστεύω θα αποτελέσει και το αντικείμενο των συνομιλιών μα σήμερα, διότι ε, δύο από τους κύριους πρωταγωνιστέ αυτού του σχεδίου επενδύσεων, ο Επίτροπο Μοσκοβισή και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Μόλτουρερ, και ο πρόεδρος της Επιτροπής των Προϋπολογισμών κ. Σαρτουή είναι εδώ παρόντες για να συζητήσουν μαζί σας. Κυρίε και κύριοι, σε κάθε πολιτική πρωτοβουλία αν έχετε ο κίνδυνος ένα ε, σχέδιο να αποτύχει όπως το σχέδιο των επενδύσεων εάν δεν ε, ανασκουμποθούμε, εάν δεν κάνουμε ο καθένας το μερίδιο της δουλειάς που του ανήκει ο κάθε ένας, η κάθε μία, η κάθε χώρα καλούμαστε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Συμβούλιο, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια, όσο και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας διαβεβαιώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο του. Τις προσεχείς εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει με μεγάλη προσοχή το σχέδιο επενδύσεων και θα υποβάλει προτάσεις και ιδέες για τη βελτίωσή του και για τρόπους ε, διασφάλισης της ε, δημοκρατικής λογοδοσίας. Η εδραίωση του σχεδίου σε μια υγεία νομική βάση είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει σήμερα να συζητήσουμε. Υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε πίσω, όπως ε, τα κριτήρια για την ε, επιλεξιμότητα των σχεδίων. Επί παραδείγματι, μια ιδέα για μια βασική, για μια βασική αρτηρία επενδυτικών σχεδίων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί, που θεωρούνται δηλαδή πιο στρατηγική σημασία, μπορεί να είναι μία λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει την πρωτοβουλία, συμμετέχει ως συνομοθέτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό σκέλος των στρατηγικών επενδύσεων. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, με τις ε, εγγυήσεις του μπορεί να δώσει τη στρατηγική διάσταση στο σχέδιο αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι η επιλογή των ε, ομιλητών μας σήμερα ιδιαίτερα σημαντική. Θα πρέπει να υποστηριχθούν τα πιο σημαντικά έργα, ε, εκείνα που θα φέρουν τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Γι' αυτό θέλουμε να ακούσουμε τις εθνικές τοποθετήσεις ε, που θα συμπληρώσουν την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευελιξία μέσα στους κανόνες, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανά, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με, μια μεγάλη, με ένα μεγάλο κίνητρο για συμμετοχή των κυβερνήσεων. Εν τέλει, η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από το ποσό της μόχλευσης και από μια ουσιαστική ρύθμιση και διευθέτηση του, κλάδου, του τομέα της διακυβέρνησης. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να ανακτήσουμε αγαπητοί φίλοι την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Την εμπιστοσύνη δηλαδή που λέει ότι μπορεί η Ευρώπη να είναι ο χώρος εκείνος, ο τόπος εκείνος στον οποίο αξίζει να επενδύουν οι ιδιώτες επενδυτές. Όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο ισχυροί. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ευρώπη έχει τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων εργασία, νέων ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Εύχομαι να έχουμε επικοδομητικές συνομιλίες και δίνω το λόγο στον αγαπητή φίλη πρόεδρο της ΣΑΕΜΑΣ, της Δημοκρατίας της Λετωνίας. Σας ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Να εκφράσω καταρχήν ε, την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Μάρτιν Σούλτζ για την ε, ε, συμμετοχή του σε πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Λετωνική Προεδρία. Ε, σήμερα εστιάζουμε την προσοχή σε ένα ευρωπαϊκό New Deal καθώς και διάφορες προβλέψεις ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προς χάρη της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι οι για τη χάρεξη πολιτικής αλλά και εμπειρογνώμονες ο καθένα στον τομέα του μετά από αρκετά χρόνια αναταραχών, στον, ελπίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπαίνει σε μια πιο ήρεμη περίοδο Ίσως η χειρότερη τρικυμία να έχει περάσει και να έχει επιστρέψει κάποια οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο η κατάσταση είναι ακόμα δύσκολη και θα πρέπει με καλό τρόπο, με έξυπνο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητές μας για να προλάβουμε τέτοιου είδους κρίσεις στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σαφές όραμα για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα για την κινητοποίηση των ιδιωτική αλλά και του ε, δημόσιου τομέα για την ε, παροχή ανάπτυξη, αλλά και για την παροχή όθησης για ανάπτυξη. Μια λεπτή ισορροπία θα πρέπει να εξευρεθεί ανάμεσα στην ε, δημοσιονομικό τομέα αλλά και τις επενδύσεις. Θα πρέπει να συνεργαστούμε ε, για να μπορέσουμε με αρμονικό τρόπο να προχωρήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να σκεφτεί το μέλλον της ε, και την ανταγωνιστικότητα, την ανταγωνιστικότητά της στον κόσμο. Θα πρέπει να βρει μοναδικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες αλλά και περιφέρειες στον κόσμο, ηλικιωμένος πληθυσμός, ε, μακριές αλυσίδες αξίας παγκόσμια, ενώ θα πρέπει να συντηρήσει τις βασικές της αξίες που περιλαμβάνουν την αλληλεγγύη καθώς και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Αυτό το νέο deal, η νέα αυτή συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει και να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις πτυχές. Οι περισσότερες επενδύσεις στην κοινωνία μας, στην παιδεία, στην τεχνολογία, στις υποδομές και η παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στους απλούς πολίτες θα οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική, αποδοτική και δυναμική οικονομία πιστεύω πως οι καρποί της οικονομικής οριμότητας, δεξιότητες, ε, κατάρτιση και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού προωθούν μεγαλύτερη αίσθηση της δικαιοσύνη στην κοινωνία. Αυτά τα βήματα είναι ουσιώδη ώστε να ε, παρεμποδιστούν οι ανισότητες που οδηγούν σε οικονομική πολιτική αστάθεια. Αν αυτές οι εναλλακτικές εφαρμοστούν, οι θεσμικές ρυθμίσεις μέσω των οποίων λαμβάνονται αποφάσεις θα πρέπει να αλλάξουν. Είναι απαραίτητο να μην υποκύψουμε στο φετιχισμό του ΑΕΠ που συχνά ε, παρεμποδίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη ή κρύβει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, Ζούμε σε έναν κόσμο με πολλούς άνεργους, πολλοί εκ των οποίων είναι νέοι και θεωρούν ότι έχουν παραμεριστεί. Ε, δεν φαίνεται να λαμβάνουμε αρκετά υπόψη την κοινωνική διάσταση ως σημαντικό στοιχείο της οικονομικής διακυβέρνησης και του συντονισμού. Αυτό είναι και το θέμα της ε, τελευταίας ε, ολομέλειας και νομίζω πως μιλώ εξ ονόματος όλων όταν λέω πως απότερο στόχος της οικονομικής μας πολιτικής είναι η ευημερία της κοινωνίας μας. Ε, η οικονομία και τα δημοσιονομικά προβλήματα οδήγησαν σε επιδείνωση των δυνατοτήτων του κόσμου να ενεργήσει, να αποφύγει την εμβάθυνση της κρίσης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν συλλογικές λύσεις όπως η πληρωμή των φόρων ή η οι κοινωνικη κοινωνικές ε, επιχειρήσεις έναντι των ιδιωτικών. Θα πρέπει το, η σφραγίδα της Ευρώπης να μπει σε ολόκληρη την κοινωνία και να εξασφαλίσουμε ότι οι πιο ευαίσθητοι, οι πιο ευάλωτοι θα μείνουν πίσω. Αν συνεργαστούμε, πιστεύω που μπορούμε να επιτύχουμε κοινωνίες πιο σύμφωνες με τις ε, θεμελιώδεις μας αρχές, ε, υπάρχουν, να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, ισχυρότερη δημοκρατία και υψηλότερε προδιαγραφές ζωής ε, διαβίωσης για ολόκληρο τον πληθυσμό μέσω των εκπροσώπων Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ένας τρόπος για τους πολίτες να ε, συμμετέχουν δημοκρατικά στην λήψη αποφάσεων. Ενώ η οικονομική διακυβέρνηση είναι περίπλοκο ζήτημα, οι εκπρόσωποι των λαών έχουν το καθήκον να διαβιβάζουν και να ε, εξηγούν τα όσα συμβαίνουν με κατανοητό τρόπο, ώστε να πείσουν τον κόσμο ε, και να έχουν την υποστήριξή του. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει τη δέσμευσή της για μια νέα συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, όπου σημαντικές πρωτοβουλίες ή προτάσεις θα υποβάλλονται και θα επεξηγούνται στα Εθνικά Κοινοβούλια από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω πως αυτή η διάσκεψη θα δώσει το βήμα για την ανταλλαγή ιδεών σε σχέση με αυτά τα θέματα. Ε, επίσης ε, να χρησιμεύσει ως έμπνευση στην αναζήτηση και την εξέβρεση νέων λύσεων μέσω της ε, ανταλλαγής εμπειριών, είτε αυτές είναι θετικές ή αρνητικές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, τώρα... Ξεκινούμε τις ε, συζητήσεις. Πρώτος λαμβάνει το λόγο ο Επίτροπος για τα οικονομικά, δημοσιονομικά, φορολογία και τελωνία. Κύριος Μοσκοβισή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε Μάρτιν Σούλτς, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, Ευχαριστώ πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Λετωνίας που προσφέρουν αυτή την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει και να συζητήσει μαζί σας για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, όπως το παρουσίασε και ίδιος ο πρόεδρος Γιούγκερ όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Στρασβούργο πριν από λίγο καιρό. Οι επενδύσει είναι όντω η πρώτη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή αυτή μπροστά στου λαού τη Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν Σήμερα, 100 μέρες μετά ε, την ανάληψη των καθηκόντων μας, να κάνουμε κάποιον απολογισμό. Το είπατε κι εσείς, Πρόεδρε, ότι η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου που μας πέρασε παρουσίασε το επενδυτικό της πρόγραμμα, που είναι αναγκαίο για να δοθεί νέα όθηση στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και να καταπολεμήσουμε τον κίνδυνο που όλοι νιώθουμε, που ζούμε, που είναι η βάλτωση των οικονομιών μας. Ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο χαιρετίστηκε από τους περισσότερους ευρωβουλευτές, από τους υπουργούς οικονομικών αλλά και από τους ηγέτες κατών και κυβερνήσεων το Δεκέμβριο. Και εξετάστηκε βέβαια και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ποιος είναι ο στόχος του επενδυτικού αυτού πακέτου. Είναι η κινητοποίηση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία προκειμένου να δοθεί νέα όθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Θέλουμε να δώσουμε μια συνολική απάντηση στις αδυναμίες που αντιμετώπισαν οι επενδύσεις και για να πάμε απευθεία στο στόχο μας, το επενδυτικό αυτό σχέδιο δεν δίνει μόνο οικονομικά μέσα, αλλά έχει και τρία επιπλέον σκέλη. Το ένα είναι η κινητοποίηση 315 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον για τις επενδύσεις για την περίοδο 2015 με 2017, ώστε να χρησιμοποιούν όσο γίνεται καλύτερα δημόσιοι πόροι που θα ελευθερώσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Στόχος μας είναι λοιπόν να χρησιμοποιηθούν καλά τα κονδύλια αυτά, κινητοποιώντας νέα μέσα, νέα εργαλεία, χρησιμοποιώντας την ε, πραγματογνωμοσύνη βέβαια της δικιάς μας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και άλλων. Για να δημιουργηθεί το ταμείο αυτό προσφέρει εγγύηση 16 δισεκατομμυρίων ευρώ η Ευρωπαϊκή Ένωση από διαφορετικούς προϋπολογισμούς. Η εγγύηση αυτή συν τα 5 δισεκατομμύρια που δίνει η ΕΤΕ θα αποτελέσουν το βάθρο του σχεδίου αυτού, του ταμείου αυτού για να προσθεθούν άλλες επενδύσεις. Επιμένω επίση, και είναι σημαντικό για εσά που είσαστε βουλευτέ, ότι δεν θα υπάρξει καμία αρνητική συνέπεια ούτε επί του κοινοτικού προπολογισμού, ούτε επί των συνιστοσών του. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δημόσια κονδύλια διαφορετικά και να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμά του. Με τη στήριξη του Ταμείου αυτού, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, λοιπόν, μαζί θα προσφέρουν 63 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το σύνολο πιστεύουμε ότι θα είναι τα 315 δισεκατομμύρια θα κινητοποιηθούν αυτά, γιατί θα έχουμε στρατηγική σημασία σε σχέδια που θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα υπάρξει ένας καταναλυτικός παράγοντας, ενισχυτικός, για να προσελκύσουμε και άλλους πόρους από ιδιωτικά ταμεία. Η ΕΤΕ μπορεί επίσης να δώσει δάνεια μέχρι 240 δισεκατομμύρια για επενδύσεις. Φαντάζομαι ότι εκπρόσωπος θα μας τα πει αυτά. Και έτσι θα υπάρξει ισχυρή κινητοποίηση ιδιωτικών κονδυλίων. Το Ταμείο επίσης θα συμμετέχει και θα προσφέρει με 75 δισεκατομμύρια ευρώ εγγύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να χρηματοδοτηθούν εκ νέου, κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι η Επιτροπή στις 13 Ιανουαρίου παρουσίασε τον κανονισμό του Ταμείου αυτού και την δημιουργία της εγγύησης αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουν γρήγορα τα πράγματα και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε σχετικά με την προτεραιότητα αυτή και ξέρω ότι και για σας Πρόεδρε αποτελεί ένα επίγον ζήτημα, μια προτεραιότητα. Όλε οι χώρε μέλη, άμεσα ή έμεσα, μέσω των δικών τους επενδυτικών τραπεζών θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην πρωτοβουλία αυτή. Και είναι σημαντικό και το λέω αυτό στους εθνικούς βουλευτές ότι πρέπει να υπάρξει ισχυρή συμμετοχή των χωρών μελών για να ενισχυθεί αυτό το θετικό μήνυμα προς τις αγορές. Όσο περισσότερο ενδιαφέρον δείξουν οι χώρες μέλη για την πρωτοβουλία αυτή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η εμπιστοσύνη των αγορών. Και για να στηριχθεί το Ταμείο από τις χώρες μέλη, που έχει έτσι καλώς τη στήριξη της Επιτροπής στην αξιολόγηση των λογιστικών των χωρών μελών, ε, μπορούν να βοηθήσουν λοιπόν και οι χώρες είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο και θα έχουν έτσι την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ζητούμε από τον ιδιωτικό τομέα, από τους επενδυτές να στηρίξουν την πρωτοβουλία μας όσον αφορά το επενδυτικό αυτό και να συμμετάσχουν σε διάφορα επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μακροπρόθεσμα που θα έχουν τη στήριξη του στρατηγικού ταμείου, του αρχικού ή να χρηματοδοτήσουν και ατομικά σχέδια. Για να γίνει αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας η επιλογή των ε, σχεδίων που χρηματοδοτεί το ταμείο να μην ε, στηρίζονται από πολιτικούς αλλά από ε, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που να μην βασίζεται η σύνθεση τη ομάδα αυτή από την εθνικότητα ή από ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά από την οικονομική του και την κοινωνική του διάσταση να κρίνονται τα σχέδια. Δεν είναι δυνατόν να ξεχνάμε και την σωστή επιστροφή. Θα πρέπει, και δεν πρέπει μάλλον να περιμένουμε καμία επιστροφή από τα χρήματα αυτά στις χώρες μέλη. Οι επενδύσεις λοιπόν πρέπει να είναι καινοτόμε και πιστεύουμε ότι ένα επιπλέον ποσό, 40 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να κινητοποιηθεί από το 2014 μέχρι το 2020. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη διάσταση. Προβλέπουμε διάφορες στοχευμένες πρωτοβουλίες προκειμένου οι επενδύσεις αυτές να γίνουν πραγματικότητα και να αποδώσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΤΕ, οι χώρες μέλη συνεργάζονται και φαίνεται από τη συνεργασία αυτή ότι υπάρχουν πάρα πολλέ επενδύσει που μπορούν να γίνουν στι υποδομέ. Καλέ επενδύσει. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν τη χρησιμότητα και ότι οι επενδύσει αυτέ όντως θα είναι βιώσιμες, παραγωγικές και ποιότητας. Ποιες είναι? Είπαμε, το σχέδιο πρέπει να είναι στοχευμένο. Ενεργειακά δίκτυα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να διαφοροποιήσουμε την προμηθειά μας. Ε, θέλουμε ψηφιακή τεχνολογία, έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία, επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα, που συχνά πρικοδοτούνται λιγότερο πόσο θα έπρεπε σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Μεταφορές, διασυνδέσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερη κυκλοφορία, καλύτερα συστήματα ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων. Δεν πρόκειται βέβαια να χρηματοδοτήσουμε τα πάντα, αλλά θέλουμε οι επενδύσεις μας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αυριανής μας οικονομίας. Θα διπλασιάσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας για να εντοπίσουμε τα προγράμματα τα οποία θα στηρίξουμε. Η ομάδα εργασίας έχει ήδη στοχεύσει σε διάφορους κλάδους και καταγράφουμε τα προγράμματα αυτά που προτείνονται, τα εντοπίζουμε δηλαδή και σιγά σιγά θα τα Θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα κέντρο συμβουλών για επενδύσεις στην Ευρώπη που θα βοηθάει την προετοιμασία των σχεδίων αυτών και την εφαρμογή τους. Θα υπάρχει πραγματογνωμοσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννοείται, από την ΕΤΕ, από τις Εθνικές Τράπεζες Επενδύσεων και από τις αρχές που διαχειρίζονται το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Επενδύσεων. Τρίτον, θέλουμε μέτρα για να βελτιωθεί η νομική ασφάλεια και να μην υπάρχουν πια φραγμοί στι επενδύσει. Και γιατί, γιατί θέλουμε μια πιο ελκυστική Ευρώπη και για να έχει μεγαλύτερε ακόμα ε, επιπτώσει, καλύτερα αποτελέσματα ακόμα το σχέδιό μα. Η εσωτερική αγορά και οι διορθωτικέ μεταρρυθμίσει αποτελούν το εργαλείο για να το πετύχουμε αυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε σε διορθωτικέ μεταρρυθμίσει. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα και για την εσωτερική αγορά για την ολοκλήρωσή της στον τομέα των υπηρεσιών, κύρια, στον τομέα των υποδομών, αλλά και στις ψηφιακές τεχνολογίες. Να, τρεις προτεραιότητες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θέλουμε να έχουμε και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει μια ακόμα που θέλουμε να φτιάξουμε τον Τζόναθον Χιλ και είναι της ε, αγοράς κεφαλαίων. Αυτά κυρίες και κύριοι ήθελα να πω και καταλήγω με το εξή. Κατά τη γνώμη μου η επιτυχία του παιδιτικού αυτού σχεδίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Πρώτον, επιγόντως, πραγματικά επιγόντως χρειαζόμαστε νομική βάση για να δημιουργήσουμε το Ταμείο. Και εδώ βασιζόμαστε πολύ στην Λετωνική Προεδρία, σας το είπα και όταν ήμουν εκεί. Βασιζόμαστε επίσης πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να δείξουν τη θέλησή του, τη βούλησή τους όλοι για να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο να μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο αυτό. Το επενδυτικό επίση σχέδιο πρέπει να επικεντρώνεται και σε επιπλέον επενδύσεις από αυτές που έχουμε ήδη στοχεύσει. Πιο στρατηγική σημασία που χρειάζεται η Ευρώπη για να αντισταθμίσουμε το, την αδυναμία μας στις επενδύσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Και τρίτον, πρέπει να υπάρχουν κίνητρα από το επενδυτικό αυτό σχέδιο, ώστε οι ΕΤΕ, οι χώρες μέλη, οι εθνικές ε, επενδυτικές τράπεζες και ο ιδιωτικό τομέα να κινητοποιηθούν, να δώσουν, να κάνουν τις επενδύσεις αυτές. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο λοιπόν που θα προχωρήσει γρήγορα και που θα έχει σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού η Επιτροπή Τελευταίες Ευκαιρίες, ξέρετε όπως τη λέμε, δίνει τις δυνατότητες. Είμαστε επικεντρωμένοι στα αποτελέσματα, σε απτά αποτελέσματα που θα έχει το σχέδιό μας αυτό το επενδυτικό στην απασχόληση, στην πραγματική οικονομία. Θέλουμε να αλλάξουμε την φυσιογνωμία, το περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Θέλουμε διαφάνεια επίσης όσον αφορά τις πληροφορίες, καλή προετοιμασία των ε, επενδυτικών σχεδίων για να επιλέγουμε βιώσιμα σχέδια και ποιότητας. Θα συνεχίσουμε, όπως είπα πριν, και τις ε, μεταρρυθμίσεις. Θα ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στα πλαίσια του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου. Φέτος, ξέρετε ότι υπάρχει η εφαρμογή, αλλά υπάρχει βέβαια και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν δεν διακόπτονται. Τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες θα συνεχίσουμε και η σημερινή συνάντηση σίγουρα είναι ένα καλό σημείο κίνησης και θέλω να πω στους βουλευτές που είναι εδώ παρόντες ότι στοιχείο κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος αυτού είναι επιπλέον σχέδια, επιπλέον επενδύσεις, καλό επενδυτικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δουλέψει σκληρά για να πετύχουμε, αλλά χρειαζόμαστε και τη βοήθεια όλων των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κύριος Μόλτσερερ, χωρίς μικρόφωνο. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Κύρια Πρόεδρε του Λετωνικού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι βουλευτέ, είναι ιδιαίτερη τιμή που αισθάνομαι να βρίσκομαι εδώ ενώπιον σα για να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δική σα τράπεζα, τράπεζα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η μετοχή τη είναι τα ε, κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να συζητήσω μέσα του εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων πάνω απ' όλα, διότι η επαφή ή άλλη η συζήτηση με τα κοινοβούλια, βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, κέριο στοιχείο της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σας χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας σε αυτή μας την ε, προσπάθεια. Κύριε Πρόεδρε, μαζί με τους συναδέλφους νομίζω εντοπίσατε το κατάλληλο θέμα συζήτησης για την ε, διάσκεψή σας. Επενδύσεις. Τα πάντα είναι επενδύσει, αλλά δεν είναι μόνο επενδύσει. Οι επενδύσει είναι μία από τι κέρυε προκλήσει. αλλά αυτέ τι κέρυε προκλήσει, αυτή την κέρια πρόκληση πρέπει να τη δούμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και από την εμπειρία μα, την εμπειρία που έχουμε από την αγορά, μπορούμε να σας περιγράψουμε μια σειρά από τις άλλες προκλήσεις. Επί παραδείγμα, τη συνέχιση της εξυγίανσης των δημοσιονομικών. Επί παραδείγμα, τη συνέχιση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς επί παραδείγματι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο επίπεδο των κρατών μελών. Κυρίε και κύριοι, τελικά πρέπει να απαλληφθούν εμπόδια και φραγμοί στις επενδύσεις που μερικές φορές, αυτό που μερικές φορές ονομάζουμε καλύτερη νομοθεσία, better regulation, το ανέφερε ήδη ο Επίτροπος Μοσκοβισή και αυτό αφορά όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη-μέλη. Και βέβαια εν τέλει πρόκληση είναι η ενίσχυση, η όθηση για τις ίδιες τις επενδύσεις. Γιατί, γιατί οι επενδύσεις είναι ο μοχλός της ανάπτυξης, μπορεί να επιταχύνει το δυναμικό ανάπτυξης. Ε, οι επενδύσεις βασικά είναι η εκ των όνου προϋπόθεση για την ενίσχυση του επίπεδου της απασχόλησης. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα επίπεδο επενδύσεων το οποίο είναι κάπως προβληματικό με την έννοια ότι είναι 15% κατώτερο από το επίπεδο πριν από την κρίση. Σε ορισμένες δε χώρες το επίπεδο συνολικά δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων είναι κατώτερο του ανώτατου επίπεδου που είχε φτάσει το 2007 κατά 50%. Θα σας δώσω κάποια επιγραμματικά στοιχεία για να σας δείξω σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και πόσο ευρύ είναι το πρόβλημα. Ξέρετε ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για το έλλειμμα το 3%. Είμαστε στο 2% αυτή τη στιγμή για, τον για τον πληθωρισμό. Συγγνώμη. Τώρα είμαστε στο 2%. Χρειάζονται για να φτάσουμε στο 3% επενδύσεις περί τα 300 30 δισεκατομμύρια, 330 δισεκατομμύρια για την έρευνα και τεχνολογία θα χρειαστούν για να φτάσουμε στο επίπεδο που έχει ορίσει ω στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την έρευνα και τεχνολογία το 3%. Επίσης για, για το ψηφιακό θεματολόγιο χρειάζονται 55 δισεκατομμύρια ευρώ ή ε, αν φτάσουμε στο ανώτατο επίπεδο που θα θέλαμε για την ε, εξυπηρέτηση των αναγκών για την παιδεία, θα μιλούσαμε τότε για 10 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ανάγκες επενδύσεων. Αυτή η απουσία επενδύσεων αποβαίνει εις βάρος και της ανάπτυξης και της απασχόλησης και εξηγεί γιατί η ανάκαμψη παραμένει σημαντικό και η πρόκληση για όλους μας. Γιατί όμως είναι μειωμένες οι επενδύσεις. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα το οποίο, στο οποίο θα πρέπει να ενσκύψουμε και να το μελετήσουμε πολύ προσεκτικά. Αυτό που γνωρίζουμε από τις αγορές, αυτό που γνωρίζουμε από τους επενδυτές είναι ότι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους δεν εκδηλώνονται επενδυτικέ ε, δράσεις είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη και ότι είναι αβέβαιο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έλλειψη εμπιστοσύνη λοιπόν, ανησυχία ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, συνδυάζονται και με λοιπά προβλήματα όπως ο κερματισμένος χαρακτήρας της αγοράς που παραμένει ισχυρό σε ορισμένα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για ορισμένα κράτη-μέλη η απλή απουσία δυνατότητας για την παρασκευή βιώσιμων σχεδίων ε, στην προπαρασκευή αλλά και στη δημοσιονομική τους εκτέλεση και ταυτόχρονα το δημοσιονομικό πλαίσιο και η ρυθμιστική ανταπόκριση στην οικονομική κρίση έχουν σημαντικά περιορίσει τις επιλογές των κρατών μελών και τις δυνατότητες που μπορεί να έχουν οι εμπορικές τράπεζες οι τράπεζες επενδύσεων ούτως Άρα λοιπόν πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, διαφορετικά θα μείνουμε πολύ πίσω. Άρα η κύρια πρόκληση για μας είναι να βρούμε έναν ευφυή τρόπο να αξιοποιήσουμε δημόσιους πόρους για να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές και να, απο... να απελευθερώσουμε το δυναμικό των επενδύσεων δεν πρέπει να βλέπουμε το δημόσιο αυτό χρήμα σαν χρήμα που θα καταναλωθεί απλώ. Θα πρέπει να το δούμε, κυρίε και κύριοι, ω παραγωγική επένδυση για την έρευνα και την ανάπτυξη, για την παιδεία. Πρέπει να το σχεδιάσουμε, να σχεδιάσουμε τη χρήση του χρήματο αυτού, κατά τρόπον ώστε να απελευθερώσει και να προσελκύσει και ιδιωτικό χρήμα επενδυτικό. Άρα λοιπόν, για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, πρέπει να αλλάξουμε πορεία και θεώρηση. Να μην μιλούμε μόνο για επιδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά για απόδοση επενδύσεων. Αλλάζουμε δηλαδή επιλογές και πορεία σε σχέση με το 1958. Θα ήθελα να εκφράσω δε τη χαρά μου για τα όσα είπε ο Επίτροπο Μοσκοβισή και για την ευκαιρία να συνεργαστούμε καλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό μήνυμα για το πώ θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να συνεργάζονται μεταξύ του. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από το 2008, από την αρχή τη κρίση, έδειξε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση με αύξηση κεφαλαίου το 2013 και μέχρι σήμερα και έχουμε ε, από τα κράτη-μέλη επιπλέον 10 δις ευρώ που κατεβλήθησαν στην, Ευρω... ΕΤΕ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είμαστε ήδη έτοιμοι να πούμε ότι είμαστε σε θέση να παραγάγουμε, να δώσουμε αποτελέσματα όπως το έχουμε ήδη πράξει. Από τα 10 δις μπορούμε να αποδεσμεύσουμε 108 συνολικά δις ευρώ. Έχουμε υλοποιήσει το πρόγραμμά μας όπως το είχαμε προβλέψει και μπορούμε σε πολύ στο χρονικό διάστημα να αποδείξουμε ότι αυτά τα 10 δις που έχουν καταβάλει τα κρατη μπορούν πραγματικά να φέρουν καρπούς. Σας δώσω μερικές πληροφορίες. Έχουμε ε, πολλαπλασιαστική λειτουργία, μόχλευση δηλαδή 1 στο 18, τα 10 δισεκατομμύρια αποδεσμεύουν 108 δις σε επενδύσεις. Έχουμε υψιστό ε, επίπεδο επιδόσεων ως προς τη μόχλευση και την παραγωγική χρήση των επενδύσεων και νομίζω ότι είμαστε σε θέση αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να το τρέξουμε, να το λειτουργήσουμε. Έχουμε εγγυημένο όγκο 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, ε, εγγύηση που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξασφαλίσει συμπληρωματική χρηματοδότηση και να προχωρήσει σε εγγραφή και υψηλότερου κενδύνου στα βιβλία της. Γιατί, Γιατί αυτή η εγγύηση με το Ταμείο σημαίνει ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις δραστηριότητες μας. Προσμένουμε ότι θα έχουμε ε, μόχλευση της τάξης του 15, 1 προς 15, με πολύ συντηρητική εκτίμηση γιατί σας εξήγησα νωρίτερα ότι τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε πολλαπλασιαστεί 18, μόχλευση ένα προς 18. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στην κατεπίγουσα ανάγκη για δράση. Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικό και εμείς να ξέρουμε πολύ νωρί ποια θα είναι τα νομικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά των κειμένων, αλλά ταυτόχρονα και να ξεκινήσουμε και να εγγράψουμε αυτή τη δραστηριότητα έστω και πριν ακόμη να τεθεί σε, εφαρμογή, σε ισχύ η νομοθεσία. Και τι σημαίνουν αυτά τα 108 δις. Δύο πτυχές έχουμε οικονομικά. Αφενός μεν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θηγατρική μας μπορεί από τα 21 δις να αφιερώσει τα 5 δις ειδικά για ένα παράθυρο που θα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις startups, για τις ε, νέες επιχειρήσεις μέχρι και τις mid caps, εκείνες που θα έχουν ανάγκη από καινοτομία και ανανέωση και άρα μπορεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με τον τρόπο αυτό να βελτιώσει την ε, παροχή κινήτρων στον όγκο των επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 75 δις για τα επόμενα τρία χρόνια. Το άλλο σκέλος είναι το σκέλος που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, εγκαθιδρύσει, τη δυνατότητα δηλαδή για υποστήριξη επενδύσεων υποδομών και καινοτομία. Ε, με τα 16 υπόλοιπα δις που καλύπτουν αυτό το σκέλος και που περιμένουμε ότι μέσω αυτών μπορούμε να δώσουμε κίνητρο για ε, άντληση επενδύσεων κατά ε, ύψους 240 δις. Αυτό αφορά μεταφορές, ενέργεια, ε, ψηφιακή τεχνολογία, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, δίκτυα, βεβαίως προϊόντα προσανατολισμένα στην κεφαλαιακή αγορά, βεβαίως προϊόντα που έχουν να κάνουν και με ίδια κεφάλαια ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μία ε, που μπορούμε και εμείς ε, να στηρίξουμε με ίδια κεφάλαια. Το δε τρίτο σκέλος, είπαμε ότι έχουμε τις μικρομεσαίες, ε, την καινοτομία και την, τις υποδομές και την παροχή συμβουλών, σαν σκέλος μπορούμε να προσφέρουμε εμείς. θα χρειαστεί και τεχνογνωσία και χρηματοοικονομική συμβουλή για τους αναδόχους, για τις δημόσιες υπηρεσίες, για το δημόσιο και τον ε, εταίρο που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι μια υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να προσφέρει τεράστιο δυναμικό ενίσχυση του δυναμικού μας. Βλέπουμε επίσης τεράστιο δυναμικό για εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις εθνικές επενδυτικές τράπεζες, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ιδιαίτερα στο επίπεδο των περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μαζί τους. Κυρίες και κύριοι, για να κλείσω. Η ΕΤΕ θεωρεί ότι το κύριο ζήτημα είναι να ανατραπεί το επενδυτικό κλίμα όπως είχε εξελιχθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Κυρίες και κύριοι, η ρευστότητα δεν αποτελεί το πρόβλημα αυτή την ε, εποχή. Η αγορά έχει ρευστότητα, έχει χρήμα, έχουν χρήμα οι αγορές. Το κέριο ζήτημα λοιπόν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς, πώς θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια στο ρυθμιστικό επίπεδο και, από την άλλη, πώς θα προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές που θα υποστηρίξουν αυτή τη στρατηγική μέσω του νέου μέσου, του νέου ταμείου. Πρόκειται για ένα νέο ταμείο, μια νέα προσέγγιση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο δηλαδή Στρατηγικών Επενδύσεων είναι μια νέα προσέγγιση που αποτελεί καινοτομία αυτό καθεαυτό το ταμείο. Ένα καταπληκτικό σύμβολο για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ενωμένη και προς το βέλτιστο συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης, των Ευρωπαίων. Χρειάζεται να ενώσουμε όλοι τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε την, την, ε, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μόλτερερ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Αρτφή. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό New Deal. Το σχέδιο που μας προτείνει η Κομισιόν με πρόεδρο τον Ζαν Κλοντ Juncker αποτελεί απάντηση στην ε, κρίση που διατρέχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτυχία του εξαρτάται από την απόλυτο συντονισμό των δράσεων και την ε, δέσμευσή μας. Καταρχήν, ο τίτλος New Deal κάνει, προκαλεί όνειρα και προσδοκίες. Ε, σημαίνει καταρχήν το να ε, καταμετρηθούν τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν και να μην κάνουμε τα πράγματα μισά. Η επιτυχία ενός πακέτου μεταρρυθμίσεων ε, μεγάλης κλίμακας του Πρόεδρου Ρούσβελτ που έβγαλε την Αμερική από την τον οικονομικό ύπνο μετρήθηκε ως μια πολιτική απάντηση που ανήρχεται στις ε, προκλήσεις ε, ιστορικά έχουμε ε, τραπεζική κρίση, μεγάλη ενεργεία, το φάσμα του αποπληθωρισμού, όμως ε, αυτό το New Deal ριζικά αντίθετα ήταν σε σχέση με το επικρατών σύστημα εδώ. Ο πρόεδρος Ρούσβελτ το πρότεινε σε ένα κογκρέσο το οποίο μπόρεσε να το υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα ανόρθωσης της οικονομίας δημόσια διακυβέρνηση των ΗΠΑ μπόρεσε να αποφασίσει, ενώ η δική μας διακυβέρνηση των Ευρωπαίων δεν ξέρουμε αν είναι στο ίδιο επίπεδο. Σίγουρα έχουμε κάποια ε, περιθώρια προόδου εδώ. Ε, τα προβλήματα της Ευρωζώνης ε, είναι συνέπεια της έλλειψης ε, διακυβέρνησης αλλά και της χαλαρότητας που επεκράτησε. Για μια δεκαετία το ευρώ σαν να είχε αναισθητοποιήσει τους πάντες συμπεριλαμβανομένων των αγορών και των ιδρυμάτων αξιολόγησης. Άρθρο 13 του συμφώνου, του Δημοσιονομικού Συμφώνου, με εντυπωσίασε γιατί ως Ευρωβουλευτής ε, συμμετείχα παλιότερα στην ε, εκπόνηση αυτού του συμφώνου και παραμένω έτσι κάπως ε, με απορία. Συζητούμε, ε, αλλά τι αποφασίζουμε τι, ποιον ελέγχουμε και τι ψηφίζουμε. θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε αυτή η διάσκεψη να είναι χρήσιμη και επικοδομητική, να εξασφαλίσει τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και τη δημοκρατική της νομιμότητα, διότι οφείλουμε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μα εποπτείας του εκτελεστικού. Είναι ευχάριστο να βρισκόμαστε μεταξύ βουλευτών, όπως είναι καθησυχαστικό να, να έχουμε το ίδιο νόμισμα, το ίδιο επιτόκιο όταν επικρατεί ηρεμία, αλλά όταν αρχίζει η τρικυμία στην Ευρωζώνη και κατά συνέπεια η στιγμή να αποφασίσουμε να κυβερνήσουμε, προς ποιον πρέπει να στραφούν οι πολίτες, από ποιον θα διζητήσουν λογαριασμό και ο κατάλογος των φορέων είναι μακρύς. Είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ο Προμόδιος Επίτροπος άμεσα ή έμεσα, είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Οικονομικής Σταθερότητας ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, είναι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων γιατί έχουν προκύψει διάφορα νέα μέσα. Εχθές το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Δημοσιονομικής Σταθερότητας, μετά ο Μηχανισμός Σταθερότητας, σήμερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και για τα δύο πρώτα ε, ε, που τα οποία σχεδιάστηκαν για να αμοιβοποιηθούν τα υπερβολικά χρέη. Στην πραγματικότητα δεν προβλέπεται κανένας ε, έλεγχος από το Ευρωκοινοβούλιο. Ας μεριμνήσουμε ώστε ε, το τελευταίο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επιδίσεων, να μην ε, ξεφύγει και αυτό από τον έλεγχο των δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων και να μην μείνει μόνο στην ΕΤΕΠ, της οποίας δεν αμφισβητώ την εμπειρογνωμοσύνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση είναι κατακαιρματισμένη και πολύ λίγο αποτελεσματική. Η διακυβέρνηση είναι ένα πέπλο ντροπή που, που, πετάμε πάνω στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αλλά και το χρησιμοποιούμε όταν δεν ξέρουμε ποιος και τι κάνει. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε μια πραγματική κυβέρνηση. Εχθές το πρωί ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ στην έναρξη της διασκεψής μας είπε πράγματα που πολλά υπόσχονται και που σηματοδοτούν νομίζω ένα καθοριστικό ε, μια καθοριστική φάση. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει κοινοβουλευτική εποπτεία σε κάθε βήμα και μόνο έτσι οι κοινοβουλευτικέ μα συναντήσει θα βρουν το νόημά του. Δεν υπάρχει ισχυρή κοινοβουλευτική δύναμη χωρί εκτελεστικό ε, το οποίο ε, να προβαίνει σε έλεγχο του, το οποίο να ελέγχεται μάλλον από το, τα κοινοβούλια. Το ευρώ που είναι η τελευταία παροχή κυριαρχίας που δεν μπορέσαμε ακόμα να έχουμε όμως δημοκρατική κυβέρνηση δημιουργεί απορίες στους συμπολίτε μας. Ωστόσο, καταλάβαμε καλά ότι όταν ε, γίνεται σεισμός, ο κίνδυνος ε, αδυναμίας πληρωμών ε, στην Ευρωζώνη, τότε τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωζώνης πρέπει να εγκρίνουν τα απαραίτητα κονδύλια. Η κρίση αυτή που διανύουμε δεν είναι οικονομική, είναι κυρίως ε, πολιτική και μόνο μέσω της πολιτικής Ευρώπης θα βρούμε τον δρόμο της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η Ευρώπη δεν θα βγει από την κρίση παρά μόνο προς τα πάνω και γι' αυτό συντρέχουν οι προϋποθέσεις νέο, New Deal. Αυτό σημαίνει νέα κατάσταση, νέα ανακατανομή των χαρτιών με τις ε, ευρωεκλογέ του τελευταίου Μαΐου, ε, τα ζάρια, ο κύβος μάλλον ερήφθη ε, και έχουμε ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μας και έναν σημαντικό ρόλο έχουμε έναν μόνιμο πρόεδρο και έτσι ε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πόληση μίξ το οποίο θα είναι υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ο σεβασμός του συμφώνου της σταθερότητας και της ανάπτυξης αλλά και ο σεβασμός του ευρώ ε, είναι απαραίτητος. Όμως η οικονομική πολιτική είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε έναν ρόλο, αυτό το ρόλο για τον πρόεδρο του Eurogroup. Τα όσα μας, μας συγκεντρώνουν σήμερα, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, άρθρο 13 αλλά και το άρθρο 16 που έχουμε, για τον ορίζοντα 2017, νέα αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνθήκων ε, προβλέπεται τότε, αλλά νομίζω πως κάτι τέτοιο χρειάζεται για να φύγουν οι ασάφειες θα πρέπει να δημιουργηθεί ίσως μια πραγματική κυβέρνηση της Ευρωζώνης με έναν πλήρους απασχόλησης ε, πρόεδρο, με πραγματικό Υπουργό Οικονομικών και τότε μόνο εμείς οι, Ευρω... οι Ευρωβουλευτές αλλά και τα Ευρωκοινοβούλια, το Ευρωκοινοβούλιο μαζί να βρίσκονται στις καλύτερες συνθήκες ώστε να μπορούν να πιέσουν τις αντίστοιχες τους κυβερνήσεις για να τροποποιήσουν το, το, το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων. Θα πληρούνται τότε οι προϋποθέσεις για να εφαρμόσουμε ένα ευρωπαϊκό New Deal με δημοκρατικό ε, δημοκρατική νομιμότητα και έτσι θα μπορέσει να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στα θεσμικά τους όργανα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Αρτσουή. Και τώρα ξεκινάει η συζήτηση. επί των τοποθετήσεων. Να σας επαναλάβω λίγο τους κανόνες που συμφωνήσαμε χθε. Έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο ομιλητών που ζήτησαν να τοποθετηθούν σε σχέση με τις παρεμβάσεις ή να κάνουν γενικές παρατηρήσεις ενδεχομένως. θα ακούσουμε τρεις ομιλητές από εθνικά κοινοβούλια και έναν ή μία βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκ με βάση βέβαια την ε, ε, προτεραιότητα κατά την οποία ζητήσατε το λόγο, θα δίνουμε το λόγο. Τώρα έχω πολύ μακροσκελή κατάλογο και γι' αυτό θα προτείνω να περιοριστούμε ο καθένας σε δύο λεπτά ερώτησης και τοποθέτησης, ώστε να έχουμε στο δυνατόν και πιο πολλές απαντήσεις από τους ε, εδώ παρόντες στο Προεδρείο. Θα κάνουμε δύο γύρους των τεσσάρων ερωτήσεων και μετά θα δίνουμε το λόγο για τις απαντήσεις, εάν συμφωνείτε. Αφού δεν βλέπω λοιπόν αντιρρήσεις, προχωρούμε έτσι και δίνω το λόγο στον κύριο Κάλεμενς από Εσθονία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σχολιάσω τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το της. Είμαι αρμόδιος για αυτά τα θέματα στο Εστονικό Κοινοβούλιο. Όλοι η Ρεν χτες είπε ότι για 40 χρόνια η Φιλανδία είναι σε ύφεση. Είναι επίσης γνωστό ότι η Φιλανδία έχει πάρει διάφορα μέτρα στην ε, εκπαίδευση για παράδειγμα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή θέση όσον αφορά την έκθεση. Οι δαπάνε της για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι 3,3%. Η διακυβέρνηση είναι αποτελεσματική κτλ. Παρ' όλα αυτά, μια τέτοια οικονομία δεν προσελκύει αρκετέ επενδύσει ούτε δημιουργεί απασχόληση. Αυτό μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε. Τι νόημα έχουν οι στόχοι του 2020. Εγώ προτείνω, κύριε Μοσκοβισή, το προσωπικό σας θα πρέπει να κάνει μια καλύτερη ανάλυση των μέτρων που προτείνετε, των στόχων δηλαδή του 2020. Κάτι λείπει. Κάτι που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, που είναι όμως βασικό για τις επενδύσεις. Και αυτό είναι το πνεύμα του επιχειρίζεστε. Η ελευθερία να είναι κανείς επιχειρηματίας, να μην έχει να υφίσταται ένα σωρό περίπλοκους κανονισμούς. Να... Το να είναι κάποιος εκατομμυρίουχος δεν σημαίνει ότι πρέπει αμέσως να πέφτει στα δόντια της φορολογίας. Από μόνο του δηλαδή δεν είναι κακό γιατί προσφέρει πράγματα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους δισεκατομμυρίχους μας γιατί τότε δεν θα έχουμε Bill Gates ε, και άλλους στην Ευρώπη αν δεν το κάνουμε αυτό. Και δεν θα έχουμε τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται εκεί όπου υπάρχουν αυτοί. ό,τι εγγύσεις δημόσιες και αν θέλουμε να δώσουμε δεν θα τα καταφέρουμε. Στην Εστονία λοιπόν αρχίζουμε το Skype, το TransferWise, διάφορες επιχειρήσεις με ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική ε, φορολογία, ηλεκτρονική ψηφοφορία κλπ. κλπ. Το πνεύμα επιχειρίζεστε δηλαδή, εμείς στην Εστονία δεν το καταπιέζουμε. Ευχαριστώ κύριε Κάλεμετς. Από την ε, Λιθουανία, ο κύριος Πούβιλατς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω ότι εμείς λέμε ότι ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια. Θέλω να επεκτείνω λιγάκι αυτή την ε, έκφραση, αυτή την ιδέα και να προσθέσω ότι οι μικροί διάβολοι κρύβονται στις λεπτομέρειες. Είναι μια φιλοσοφική ρίσκη. Η φιλοσοφία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο φασισμός είναι παραδείγματα καταστροφής ολόκληρων εθνών και τάξεων. Αν έχουμε μια καλή φιλοσοφία, καταλαβαίνουμε καλύτερα την κατεύθυνση και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Με τη φιλοσοφία μπορούμε να προχωρήσουμε σωστά. Είναι ένα δημόσιο αγαθό η φιλοσοφία. Συζητώντας λοιπόν για New Deal, νέα συμφωνία, θα έπρεπε να ξαναδούμε τις απόψεις μας όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κατά τη γνώμη μου, ατομικισμός ή νεοφιλελευθερισμός είναι αυτά που κυριαρχούν σήμερα στον κόσμο. Και αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Εμείς υποτιμούμε το μηχανισμό της αλληλεγγύης, του κοινού αγαθού και άλλα τέτοια πράγματα. Θέλω όμως να μας υπενθυμίσω ότι εμείς οι πολιτικοί είμαστε για να εξυπηρετούμε το κοινό, τον κόσμο, το δημόσιο αγαθό, όχι το ιδιωτικό. Μια ολιστική λοιπόν άποψη απέναντι στο New Deal, την αυτή συμφωνία, θα έπρεπε να είναι και το αντικείμενο των μελλοντικών μας συζητήσεων. Ευχαριστώ. κύριος από την Γερμανική Βουλή, Bundestag. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το New Deal είναι ένα μεγάλο ιστορικό υπόδειγμα και παράδειγμα. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα λοιπόν αυτή η ευκαιρία που μας προσφέρεται με το επενδυτικό πακέτο δεν πρέπει να χαθεί με έστω και δικαιολογημένες επιφυλάξεις για ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα εθνικά κοινοβούλια, είτε τη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, είτε το ευρωπαϊκό, δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν με τι επιφυλάξει του ε, αυτό το σχέδιο και την αποδοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιτύχει αυτό το σχέδιο το επενδυτικό. Πρέπει ο πολίτης να διαισθανθεί ότι η οικονομική και η κοινωνική πραγματικότητα θα βελτιωθούν σημαντικά. Μία βεβαιότητα την οποία δυστυχώ δεν βλέπουμε σε πολλά μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει με ιδιαίτερη προσπάθεια να υποστηρίξουμε για να αλλάξει ροή ο ποταμό. Πρέπει λοιπόν χρόνια τώρα που έρχομαι εδώ στις Βρυξέλλες, γιατί και πέρσι ήμουν εδώ, να σταματήσουμε να κάνουμε ε, επιφανειακές ιδεολογικά προσανατολισμένες μόνο συζητήσεις. Πρέπει να την ξεπεράσουμε αυτή τη συζήτηση και να επιδιώξουμε έναν ουσιαστικό στόχο. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο μπορεί να μας κινήσει για να δείξουμε στους ανθρώπους ότι πραγματοποιούμε πρακτικά βήματα για την αλλαγή στη ζωή τους. Στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερμανία, γιατί και στη Γερμανία πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά και να προχωρήσουμε σε μεγάλες επενδύσεις. Είναι τεράστια η ευκαιρία που προσφέρεται, είναι ευνοϊκή η συγκυρία, έχουμε μεγάλη αδυναμία επενδυτική στην Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς το πρόγραμμα αυτό έχετε την κατάλληλη στιγμή και στην κατάλληλη θέση. Και στον κύριο Αρτσουή και τους λοιπούς που είπαν ότι υπάρχουν ακόμα ε, εκρεμή ζητήματα, όχι μόνο για εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια, αυτό θέλω να επισημάνω. Ε, το δεύτερο, μια ουδέτερη διαδικασία επιλογής, πολύ ωραία και το λέω αυτό ως εκπρόσωπο πως ενός κράτους με ισχυρή οικονομία και ανάπτυξη, όπως ονομάζεται τουλάχιστον. Πρέπει να φροντίσουμε η, ε, το χάσμα, η τάφρος μεταξύ των πιο ευημερούντων και των οικονομικά λιγότερο στεναρών κρατών να μην ενισχυθεί, να μην αυξηθεί το χάσμα αυτό εξαιτία του προγράμματος. Όπω είπα, η αλλαγή κλίματο θα μπορέσει να προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα πολλά από αυτά που υπόθηκαν τι τελευταίε μέρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το Βασικότερο στόχο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη είναι να φτάσουν σε μια ισορροπία και να φτάσουν σε χρέο λιγότερο του 3% του ΑΕΠ. Τώρα οι επιμονωμένε κυβερνήσει θα πρέπει να αποφασίσουν πώ θα φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, υποτίθεται ότι αυτό γίνεται με τη, επί τη βάση των ε, υπολογισμών τη Eurostat, αλλά γίνεται τελικά επί τη βάση ε, του ρευστού. Ε, έχουν την ίδια μέτρηση με κάθε ευρώ που δαπανάτε για τις τρέχουσες δαπάνες. Ωστόσο είναι σαφές ότι ένα ευρώ που δαπανάτε για επένδυση έχει τελείως διαφορετική οικονομική σημασία από ένα ευρώ που δαπανάτε για κοινωνικές ε, ε, παροχές. Ως αποτέλεσμα, συμμορφούμενοι προς το σύμφωνο αυτό, οι κυβερνήσεις βρίσκουν ότι είναι πολύ πιο βολικό πολιτικά να περικόπτουν τις επενδύσεις παρά να περικόπτουν τις κοινωνικές τους ε, δαπάνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει το πρόβλημα αυτό επανειλημμένα. Εδώ και καιρό εκφράζουμε τη λύπη μας για τη μείωση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη, όπως και σήμερα το πρωί. Ίσως να μην ήταν μια μη θελημένη συνέπεια των ε, κανόνων ε, του συμφώνου, όμως όταν εφαρμόζονται τελικά, όπως είπαμε, τα κράτη ε, ενστικτοδός περικόπτουν τις επενδύσεις. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα ταμείο του Γιούνκερ για να, για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να συμμετέχουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ότι οι δαπάνες που, συμπε... συρρυκνώνονται για να γίνουν δημόσιες επενδύσεις θα αποκλειστούν από τις υπόλοιπους κανόνες ε, SGP. Η ίδια λογική θα πρέπει να εφαρμοστεί για να εξαιρούνται στην περίπτωση αύξηση δημοσίων επενδύσεων οι επενδύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη, οι εθνικές κυβερνήσεις μέσω των εθνικών τους κοινοβουλίων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Ζάντα. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Ζάουρερ από το Ισπανικό Κοινοβούλιο και αγαπητοί συνάδελφοι παρεμπιπτόντος. Ένα λεπτό κύριε Ζάουρερ. Εάν θέλετε μπορείτε να εγείρεστε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής σας. Είναι ε, συνήθεια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλωστε, διευκολύνει να σα βλέπουν οι συνάδελφοι. Εφόσον το επιθυμείτε, φυσικά. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε. Είτε να μιλήσετε καθιστή, είτε να εγερθείτε. Να, κύριε Ζάουρερ, τώρα σα φέρνω σε δύσκολη θέση. Μπορείτε να πάρετε το λόγο, λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αποτελεσματικότητα του νέου δημοσιονομικού συμφώνου πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου αλλά επιδέχεται βελτίωση η ευελιξία του συμφώνου σταθερότητας. Γιατί για λόγους οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί και έχουν σχολιαστεί πολύ, αλλά θα ήθελα να τους αναφέρω και εγώ σε αυτή την ε, ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση που έχουμε. Το πρώτο είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη παρουσία δημοσίων κεφαλαίων σε αυτό το επενδυτικό πακέτο. Διότι έτσι όλο και περισσότερα επενδυτικά σχέδια μπορούν να έχουν παρουσία στο σύνολο αυτών των ε, προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή πρέπει την ε, απόδοση του ιδιωτικού να τη συγκρίνουμε με την απόδοση του δημοσίου. Γιατί μιλάμε για την απόδοση που θα έχει μακροπρόθεσμα πολλαπλασιαστικά η οικονομία μας. Έτσι δεν είναι. Δεύτερον, πρέπει να αποκλείσουμε τις χώρες του διορθωτικού σκέλους διότι οι χώρες αυτές συνεχίζουν να εφαρμόζουν κάποιους κανόνες μεσοπρόθεσμα όταν κάνουν στρατηγικές επενδύσεις ή όταν κάνουν μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικού τύπου δεν είναι λογικό οικονομικά να του ζητήσουμε κι άλλα. Όλες οι χώρες που είναι σε αυτό το διορθωτικό σκέλος, αλλά και στο προληπτικό σκέλος, όλες αυτές έτσι κι πρέπει να βελτιώσουν την ανάπτυξη της οικονομίας τους, όλες. Γιατί λοιπόν μιλάμε για αυτές τις χώρες, γιατί να μην χρησιμοποιούνται, να μην περιλαμβάνονται και αυτές την ευελιξία την οποία θέλουμε να προσφέρουμε στις άλλες. Είναι μια χαμένη ευκαιρία. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν προκυκλικά αποτελέσματα άλλες όχι. Εμείς εδώ θέλουμε οικονομική ε, ανά... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σάουρερ. Ρόσμαν, Αυστριακό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος Ιουνκέρ είναι ένα φιλόδοξο σύνολο μέτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων. 21 δις ευρώ μόνο όμως, όχι φρέσκο χρήμα, με μόχλευση της τάξης του 15. Αυτό δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί πιστεύω. Και επιτρέψτε μου να διατυπώσω κάποια επικριτικά σχόλια σε σχέση με αυτό το επενδυτικό πακέτο. Από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει να εφαρμόζεται και θα μπορέσει ε, βραχυπρόθεσμα μόνο να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αυτό δεν θα αρκέσει για να λύσει τα προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν να δώσει βεβαίως να δοθούν δημόσιες επενδύσεις και ενίσχυση ε, κίνητρα για τις ιδιωτικέ, αλλά δεν αρκούν αυτές. Θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς τοποθετήσεις ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη αυτό δεν εξασφαλίζεται επαρκώς. Και αν επιπλέον το επενδυτικό αυτό σχέδιο είναι να αναπτύξει κάποια αποτελέσματα, αυτό, αυτά τα αποτελέσματα θα είναι μόνο αλλαγή σε σχέση με τη δυστημία που επικρατεί και τη δυσφορία. Εφορία πάντως θα θα δούμε. Το νέο, νέο deal αυτό, η νέα αυτή συμφωνία δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι. Γιατί για να είναι πραγματικό New Deal αυτή η νέα συμφωνία και το πακέτο επενδύσεων θα χρειαζόταν σχέδιο επενδυτικό, πρόγραμμα επενδυτικό που να αξίζει πραγματικά το όνομα επενδυτικό πρόγραμμα. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να είναι ένα πράσινο επενδυτικό πρόγραμμα πάνω απ' όλα ώστε να μην ενισχύονται πυρηνικές ε, μονάδες παραγωγής πυρηνικής ε, ε, ενέργειας από τα πυρηνικά χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα για ένα ουσιαστικό πυρηνικό, ένα ουσιαστικό συγγνώμη, ε, επενδυτικό πρόγραμμα. Η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού τομέα. Γιατί πάντοτε έχουμε επενδύσεις στο χρηματοοικονομικό τομέα και όχι στον πραγματικό τομέα της οικονομίας. Και γιατί δεν έχουμε υποστήριξη από το, τις δημόσιες επενδύσεις, το χρήμα του, του φορολογουμένου ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των υποδομών. Αυτές έπρεπε να είναι πάντα στο δημόσιο. Ευχαριστώ Χάρισον, Λόρδο Χάρισον, από την Βουλή των Λόρδων. Κύριε Πρόεδρε, χτες ε, η Βουλή των Λόρδων δημοσίευσε την έκθεσή της ε, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο μετά την, Ευρωπαϊ... μετά την δημοσιονομική κρίση. Ε, το έχω εδώ. Ένα κεφάλαιο αναφιερώνεται στην ε, θεματολογία της ανάπτυξης. Ε, ποιον μας ήρθε χτες ο Τζόναθαν Χίλ για να μιλήσει για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών και μάλιστα κάνουμε σεμινάριο στην Βουλή των Λόρδων την επόμενη εβδομάδα που η Σάρον και ο Τζόναθαν Φόλτ θα μιλήσουν. Ε, όμως έχω μια ερώτηση ε, στον πρώην Ευρωβουλευτή Πιέρ Μοσκοβίτσι όσον αφορά το πρόγραμμα επενδύσεων στην Ευρώπη και κατά πόσο η αναλογία του 15 προς 1 δημόσια χρήματα που υποτίθεται θα μοχλεύσουν ε, ιδιωτικά χρήματα είναι ρεαλιστική. Και αυτό ε, την ερώτηση την υποβάλλω και στον κύριο Μόρτερ από την ΕΤΕΠ. Προς τον κύριο Μασκοβίτση επίσης θέλω να απευθύνω την, την εξή παρατήρηση. Ο ενιαία αγορά είναι ο ταχύτερος δρόμος για την ανάπτυξη και την θέση απασχόληση. Αλλά υπερβολικά πολλά εθνικά κοινοβούλια αντιστέκονται. Τι μπορεί να γίνει ώστε να εξασφαλιστεί μια πραγματική αγορά 28 χωρών και και η δική μου κυβέρνηση είναι ε, ένοχη για το ίδιο. Σε έναν άλλον παλιόφιλο, τον Ζαν Αρτουή, που είναι τώρα πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ήθελα να τους ζητήσω να σχολιάσει τον προϋπολογισμό 2014-2020, το πολιτές δηλαδή, και κατά πόσο θα υπάρξει αλλαγή ώστε να κατευθυνθούν όχι απαραίτητα όλα τα χρήματα, αλλά η κατεύθυνση των χρημάτων αν θα αλλάξει προς την ανάπτυξη ε, και τέλος αυτή την έκθεση επενούμε το Ευρωκοινοβούλιο και την ε, Sharon Bowles για ο Μισελ Μπαρνιέ, επίσης ο περχόμενος ε, ε, επίτροπος επενείται, αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και τον πρόεδρο, του Χέρμαν Φαν Ρόμποϊ. Μπράβο τους. Λόρδε Χάρισον, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ιστορική στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποτέ δεν άκουσα Βρετανό εκπρόσωπο Κοινοβουλίου να μιλήσει τόσο καθαρά υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σα ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Φερέιρα τώρα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρακαλώ κυρία Φερέιρα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την Επιτροπή για το γεγονός ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Ταμείου Επενδύσεων. Αυτό αντιπροσωπεύει την αναγνώριση του ότι χρειάζεται μια νέα δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι χωρίς λίγο οξυγόνο δεν, ε, δεν θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ωστόσο θα ήθελα και κάποιες απαντήσεις. Ε, ε, ο προβληματισμός μου αφορά ακριβώς το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα της προσαρμογής που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης έγινε ε, εις βάρος ε, των ε, δημοσίων επενδύσεων, με τις περικοπές αυτών δηλαδή, για λόγους που πριν από λίγο εξήγησε κάποιος συνάδελφος. Οι επενδύσεις λοιπόν περικόπηκαν και κυρίως ε, στις χώρες όπου είναι υποπρόγραμμα για υπερβολικό χρέος, οι περικοπές αυτές ήταν κάθετες απόλυτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία ε, δυσχεραίνουν την πρόσβαση στους μηχανισμούς αυτούς. Μία είναι η ιδέα της ε, μακροαιρεσιμότητας που επιτρέπει, που μάλλον που υποχρεώνει αυτές τις χώρες σε συνέχιση αυτής της κατάστασης αν δεν τηρούν όλους τους κανόνες του συμφώνου. Ε, Επίση, ε, αυτό που είπε ο συνάδελφο Σάουερ πριν από λίγο για τους κανόνες ευελιξία, τη ρήτρα επενδύσεων και το κατά πόσο αυτή θα, θα επεκταθεί για τις χώρες που είναι σε προγράμματα. Τέτα... Τρίτο στοιχείο το οποίο μόλις επιβεβαιώθηκε είναι ότι στην ανάλυση κινδύνου επικρατεί αυτή η κουλτούρα του τομεακού κινδύνου αλλά δεν προβλέπεται τίποτα σε σχέση με την ε, έναν κίνδυνο αναχώρα. Ε, άρα λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις υπάρχουν κάποιες χώρες που θα είναι πιο ευνοϊκές για να αναλάβουν προγράμματα και να προχωρήσουν σε παιδι και να προβούν σε επενδύσεις. Και το ερώτημά μου είναι μήπως έτσι ε, επιδεινώσουμε ακόμη περισσότερο τις ανισότητες μέσα στην Ένωση εάν δεν λάβουμε υπόψη αυτές τις πτυχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φερέρα. Ακούμε πρώτα τον κύριο Μοσκοβισή, μετά τον κύριο Μόλτερερ και στο τέλος τον συναδελφό Αρτουή. Κύριε Μοστοβίσκη, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές που τοποθετήθηκαν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία. Πρώτον, θα υπενθυμίσω το σχέδιο επενδύσεων ανταποκρίνεται, αποτελεί απάντηση σε μία διάγνωση την ανεπάρκεια των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έλλειμμα επενδύσεων, τα μιλούμε για την περίοδο πριν το 2008 και μέχρι το 2014. Υπάρχει μια διαφορά 15 με 20% προς το ύψος των επενδύσεων σε σχέση με το 2008, προς τα κάτω. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε ποια είναι η πρόκληση για μας. Εάν δεχθούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει το ρόλο της ως πρώτης οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, ακριβώς εκεί που μπορούν κάποια κράτη να έχουν υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων, χάνουμε την πρωτοκαθεδρία μας και τη δυνατότητα να καθοδηγούμε, να είμαστε ηγετική δύναμη στην παγκόσμια οικονομία. Ακριβώς εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση. Πρέπει εξάπαντος αυτή την αυτό το έλλειμμα σε επενδύσεις να το απορροφήσουμε και σε αυτό θα συμβάλλει σημαντικά ουσιαστικά το σχέδιο επενδύσεων. Δεν θα είναι παρκές, το είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, θα πρέπει ίσως να το παρατείνουμε και να το διευρύνουμε εάν χρειαστεί, αν και εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματικό όπως το ελπίζω. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν για την επιχειρηματικότητα, για την εσωτερική αγορά. Εγώ είπα ότι το σχέδιο αυτό είναι κομμάτι μιας ευρύτερης προσέγγισης. Έχει τρεις, τρία σκέλη, τρεις πυλώνες αυτή η προσέγγιση επιτροπής. Τη δημοσιονομική εξυγίανση, να έχουμε γερά δημοσιονομικά. Πρέπει να μειωθούν τα ελλείμματα, είναι απαραίτητο αυτό, έστω και αν προβαίνουμε σε μια νέα ερμηνεία, πιο ευέλικτη όπως γνωρίζετε σε σχέση με ερμηνείε που είχαν δοθεί στο παρελθόν. Δεύτερον, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τίποτε δεν μπορεί να μας επιτρέψει να οπισθοδρομήσουμε σε σχέση με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο σχέση με το παρελθόν που είδαμε ότι η λιτότητα δεν φέρνει ανάπτυξη, αλλά για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Για να έχουμε μια ανοιχτή οικονομία που είναι η οικονομία μας και εδώ έρχομαι στην επιχειρηματικότητα γιατί είναι σαφές ότι η Επιτροπή αυτή, όπως και η προηγούμενη σύνθεσή της, γνωρίζουν πολύ καλά από πού προέρχεται ο πλούτος, πού παράγεται πλούτος, μέσα στην επιχείρηση παράγεται ο πλούτος και όχι σε κάποιο είδους ή προτύπου ε, κρατιστικής ή υποεποπτείαν οικονομίας. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ιδιωτική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και υποστήριξη από τις δημόσιες επενδύσεις. Και έτσι προχωρώ στην επόμενη παρατήρηση που έχει να κάνει με την ευελιξία που πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν ως μέσος, μέσον για την ενίσχυση των επενδύσεων και της, ε, την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Στις 13 νομίζω Ιανουαρίου ξεκινούμε με, μια, με ένα νέο άνοιγμα και δημιουργία χώρου ευνοϊκού για τις θετικές επενδύσεις. Εάν δηλαδή ένα κράτος θέλει να αξιοποιήσει σημαντικό ένα, κομμάτι αυτού του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για να στερεώσει την ε, αξιοπιστία του. Αυτό δεν θα υπολογιστεί ως χρέος ή ως έλλειμμα. Δεν θα το βάλει δηλαδή σε μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Αυτό ισχύει για όλα τα κράτη, ανεξαρτήτως της θέσεώς τους, ε, σε ένα διορθωτικό ή προληπτικό σκέλος του συμφώνου. Στη συγχρηματοδότηση επίσης πάλι δεν θα ε, υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο ως χρέος, ως έλλειμμα. Γιατί δεν θέλουμε κανείς να αποθαρρυνθεί και να ε, μην τολμήσει να μπει μέσα σε αυτό το σχέδιο των επενδύσεων. Θέλουμε να δώσουμε ισχυρά κίνητρα στα κράτη για επένδυση. Και εδώ απευθύνουμε στους εθνικούς βουλευτές. Αυτή είναι η επιδίωξή μας η βούλησή μας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα κράτη-μέλη, με τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν τις επενδυτικές τους τράπεζες δηλαδή, πρέπει να προχωρήσουν. Και μια τρίτη παρατήρηση, το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο ευρύ, στόχο έχει βεβαίως να ενθαρρύνει τις επενδύσεις, αλλά θέλει να τι ενθαρρύνει με τρόπο στοχευμένο. Το είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση. Δεν θα ενθαρρύνουμε, δεν θα χρηματοδοτήσουμε ή ανδήποτε επένδυση. Δεν θα κοιτάξουμε μόνο με πνεύμα την ισότιμη ανταπόδοση, την ανταπόδοση της επένδυσης. Ε, αλλά θέλουμε να έχουμε μια υποστήριξη των επενδύσεων οι οποίες θα έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, θα ενισχύσουν κάτι που ήδη γίνεται. Δεν θα ε, στηρίξουμε επενδύσεις οι οποίες ούτως ή άλλως θα γίνονταν. Θέλουμε νέες επενδύσεις οι οποίες θα έχουν οικονομικό βεβαίως όφελος να προσφέρουν, αλλά που ενδεχομένως να μην μπορούσαν να αντλήσουν χρηματοδότηση και άρα θα τους επιτρέψουμε τον τρόπο αυτό να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Αυτό έχω να πω και ίσω ο Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων να έχει να πει περισσότερα, αλλά ακριβώ αυτό μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κλείνω, Πρόεδρε. Ότι η ΕΤΕ είναι μια τράπεζα με τριπλό Α. Μπορούμε να τη βοηθήσουμε λοιπόν να επενδύει περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Το είχαμε πει και στο παρελθόν με τον Υπουργό Οικονομικών ε, της Γαλλίας ε, που ήμουν εγώ τότε και ο, τον κύριο Σόιμπλε, Υπουργό των Οικονομικών της Γερμανίας. Θα κοιτάξουμε και αυτούς που είναι πιο αδύναμοι στις ε, αγορές, αλλά πάνω απ' όλα θα τους δώσουμε εγγυήσει για να προχωρήσουν. Εγώ έχω κάθε εμπιστοσύνη στις τράπεζα, στην τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί είδαμε ότι έχει μόχλευση της τάξης του 18%. Άρα πρώτα αντλείται από την αγορά και πάμε στα 63 ε, δισεκατομμύρια ευρώ και μετά μπαίνει στην ε, αγορά η μόχλευση που μας φτάνει στα 200 εκατομμύρια. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε για να επιτύχει το σχέδιο αυτό μια Ευρωπαϊκή Ένωση στις διάφορες της πτυχές, θεσμικά όργανα, αλλά και τα θεσμικά όργανα και οι δημόσιες επενδυτικές τράπεζες. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω και εγώ και θα απαντήσω για τον πολλαπλασιαστή. Από όσο γνωρίζετε, η εμπειρία μας, εμπειρία που βασίζεται και στην αύξηση κεφαλαίου, τα 10 δισεκατομμύρια που αρχίσαμε το 2013, τότε περιμέναμε και υποσχεθήκαμε ότι πρόκειται για κίνητρα για 180 δισεκατομμύρια και είχαμε αποτελέσματα. Δεν έχω βέβαια ακριβώς τα ποσά για τα τέλη της χρονιάς, αλλά ο πολλαπλασιαστής είναι τουλάχιστον 1 προς 18. Αυτή είναι και η βάση. Γι' αυτό και είμαστε σίγουροι με το 1 επί 15. Αλλά όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το στοιχείο κλειδί είναι να έχουμε μια τέτοια δόμηση του ταμείου που να υπάρχει ευελιξία και να μπορούν να κάνουν πρόβλεψη ιδιωτικοί επενδυτές. Ο πολλαπλασιαστής ε, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να ξέρουμε ότι θα υπάρξουν τα δάνεια, ότι θα προστατευτεί συγχρόνω το τριπλό Α και θα έχουμε τα οικονομικά μέσα εκείνα τα οποία θα προσελκύσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις Είμαστε σίγουροι με το 1 προς 15. Πιστεύω ότι είναι προβλέψιμο, ότι είναι μια υπόθεση απόλυτα ρεαλιστική. Δεύτερον, όσον αφορά τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά. Εμείς ως ΕΤΕ θα επιλέξουμε τα προγράμματα βάσει κριτηρίων ε, τραπεζικών. Δηλαδή οικονομικά πρέπει να είναι υγιή, τεχνικά πρέπει να είναι υγιή και περιβαλλοντικά επίσης να στέκουν. Διότι είναι ένα δάνειο το οποίο εμεί δίνουμε. Οπότε τα προγράμματα πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα ε, χρήματα, απόδοση. Έπειτα, τα κράτη-μέλη θέλουμε να επενδύσουν. Εγώ αναμένω τις δεσμεύσεις των χωρών ε, μελών σε δύο επίπεδα. Σε επίπεδα προγραμμάτων ή δυνατών και δεύτερον σε επίπεδο εθνικών επενδυτικών πλατφόρμων. Γιατί εδώ οι χώρες μέλη μπορούν να έχουν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις δικές τους καταστάσεις, όπως γίνεται στη Γερμανία. Αυτό είναι θέμα δηλαδή των χωρών μελών. Πώς θα κάνουν τις επενδύσεις, αν δεν γίνουν στο Ταμείο, αλλά γίνουν στις εθνικές επενδυτικές ε, πλατφόρμες. Για την συνοχή, εδώ έχω μια απλή απάντηση. Η πρωτοβουλία Juncker έχει ως στόχο να στηρίξει την πολιτική συνοχής. Γιατί, Γιατί μπορούμε να προσελκύσουμε και να κάνουμε πιο εντατική χρήση προγραμμάτων μας όπως το Γιάσπερ στον τομέα της συνοχής. Έχουμε επεκτείνει το εύρος του Γιάσπερ όχι μόνο για τις νέες χώρες μέλη, αλλά για όλες τις περιφέρειες συνοχής. Και συγχρόνως μακροπρόθεσμα τα οικονομικά εργαλεία προσελκύουν και αυξάνουν την δυνατότητα απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων. Τέλος. Περιμένουμε τις αποφάσεις των κοινοβουλίων για να αρχίσει να ισχύει το ΕΦΣΥ το Σεπτέμβριο που μας έρχεται το επενδυτικό αυτό ταμείο. Αλλά επίγει η κατάσταση. Η ΕΤΕ μπορεί να βοηθήσει στο μεταξύ με την υπόθεση ότι θα καλυφθεί και αυτή η βοήθειά μας με τις εγγύησεις που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό έχουμε υπόψη μας. Τελευταία, πραγματικά τώρα τελευταία μου παρατήρηση. Την πρωτοβουλία Juncker μην τη βλέπετε σαν ένα ενιαίο πράγμα. Είναι μια πρωτοβουλία που καλύπτει και τις διασωτικές μεταρρυθμίσεις και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και βέβαια τη δημιουργία του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου δηλαδή Διαρθρωτικών Επενδύσεων. Ελπίζω να μην υπάρχουν πια εμπόδια στις επενδύσεις. Χρειάζεται εντατική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα κάνουμε και θέλουμε να συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την νομοθετική πρόταση. Γιατί υπάρχουν μερικά θέματα που έχουν σημασία για μας. Το θέμα της ποιότητας των εγγύσεων, για παράδειγμα. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί για να διατηρήσουμε το τριπλό μας α το θέμα των κυβερνήσεων, το θέμα της προσθετικότητας. Είναι ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε έγκαιρα σε όσο γίνεται καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε, κύριε Μόλτερερ. Κύριο Συνεχίζουμε. Με τον κύριο Αρτουά. Αρτουή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να χαιρετήσω τον Λόρδο Χάρισον. Το πιο φιλοευρωπαϊστή Βρετανό βουλευτή. Η παρουσία του μεταξύ ημών μας επιτρέπει να υπογραμμίζουμε, να υπογραμμίσουμε σε ποιο βαθμό η διάσκεψη του άρθρου 13 του Fiscal Compact είναι μια διάσκεψη σημαντική και αυτό το επισημαίνω γιατί δεν το έχει υπογράψει το Fiscal Compact το Ηνωμένο Βασίλειο και ευχαριστώ πολύ τον ε, φίλο Χάρισον για τις φιλοευρωπαϊκές του θέσεις και την υποστήριξή του. Δεύτερη παρατήρηση για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ασφαλώς ε, είναι πολύ σκληρό, ασφαλώς δεν κάνουμε αρκετές διακρίσεις μεταξύ ε, επενδύσεων και λειτουργίας. Και βλέπω ότι μπορεί η από δηλαδή μέτρα που έχουν δημοσιονομική ε, λειτουργία σε σχέση με επιχειρήσεις πιστοτικές ε, δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο. Για τις αποφάσεις και εδώ παραπέμπω στον Αλμπέρτο Γκουαλτιέρη που είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Σωματικών Υποθέσεων θα πρέπει νομίζω ιδιαίτερα να ενισχύσουμε ακούγεται διαρκώς το κινητό του ομιλητή στο μικρόφωνο ε, πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την νομική βάση και πρέπει να έχουμε αντίληψη ότι σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο προχωρεί ταχύτατα όταν λαμβάνονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμείς βρισκόμαστε σε ενός είδους αδράνεια αδράνεια η οποία μας φέρνει σε πολύ δυσμενέτερη θέση και επιδεινώνει τις συνθήκες για τις δράσεις που θέλουμε να αναλάβουμε. Θέλω λοιπόν ταχύτατα να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, με την νομική βάση και τα νομιμοθετήματα που χρειάζεται για να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να γίνει πραγματικότητα. Euh, η επιτυχία εξαρτάται από τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που θα υλοποιήσουν τα κράτη. Θέλω να το υπογραμμίσω και αυτό. Ε, πολύ αμφιβάλλω για το αν θα μπορέσει να στεφθεί με πραγματική αποτελεσματικότητα και επιτυχία το σχέδιο ε, Juncker όταν δεν έχουν υλοποιηθεί διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει όπου χρειάζονται. Βεβαίω, μικρέ και μέσε επιχειρήσει έχουν δυσκολία στη χρηματοδότησή του. Αλλά όταν εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα, εν γέννη οι επιχειρήσει εξασφαλίζουν του χρηματοοικονομικού πόρου που χρειάζονται. Άρα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να γίνουν στην κάθε χώρα. Στην κάθε χώρα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αυτό θα είναι και το τίμημα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου. Χρειάζεται ανταγωνιστικότητα για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να καμφθεί η καμπύλη της ανεργίας. Αυτές ήταν οι δικές μου παρατηρήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Αρτουή. Συνεχίζουμε. Σας παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας, όπως αποφασίστηκε από το μου. Έχουμε τρία εθνικά κοινοβούλια και μετά έναν ευρωβουλευτή. Και μετά άλλο ένα κύκλο και μετά θα απαντήσουν εδώ οι καλεσμένοι μας. Κύριε Ρερή, Ιταλία, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους ομιλητές ότι το να, να ζωπηρωθεί και να εδραιωθεί μια ισχυρή οικονομία στην Ευρωζώνη χρειάζεται ε, ε, ε, μεγάλες επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων και θα μπορούσαν έτσι να κινητοποιηθούν νέες πηγές ανάπτυξης και στην πλευρά της ζήτησης όσο και της ε, ε, παροχής. Μέσο και μακροπρόθεσμες επενδύσεις δεν είναι απλά μια χρονική ε, εφεύρεση. Θα πρέπει να θεωρηθεί στρατηγική σημασία για το μέλλον της ευρώ και της ευρωζώνης. Τούτου λεχθέντως υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να έχουμε ένα επιτυχές επενδυτικό σύμφωνο όπως αυτό που προτείνεται θα αναφέρω δύο προϋποθέσεις εξ αυτών. Καταρχήν, η το μέγεθος αυτού του νέου επενδυτικού προγράμματος θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να έχει οικονομικό αντίκτυπο. Όπως ξέρουμε, η μείωση των επενδύσεων σε ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε 350% ετησίως. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το πλάνο που αυτή τη στιγμή προτείνεται. Ακόμα και με τα πιο αισιόδοξα σενάρια θα είχαμε περίπου 100 ή 105 ετησίως. Ε, ε, ερώτησή μου λοιπόν είναι ότι πρόκειται για μια e e, ένα e ευφυές επενδυτικό πρόγραμμα από οικονομικής άποψης, αλλά σε πρακτικούς όρους υπάρχει μέγας κίνδυνος ότι από αυτή τη μορφή δεν θα λειτουργήσει ως οικονομική όθηση. Δεύτερον, Συμφωνώ απόλυτα πως είναι πολύ σημαντικό, σημαντική μια τεχνική, τεχνικός έλεγχος, μια προεπιλογή των επενδύσεων, δηλαδή σε τεχνικό επίπεδο. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικό πλάνο, μια γενική πολιτική, οικονομική, στρατηγική και αυτή τη στρατηγική δεν τη διακρίνω. Ε, πώς, πώς εμφυλιώνουμε το επενδυτικό μας προγράμματα με τα υπόλοιπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι θα πρέπει επίσης να επιλέγονται σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Τεχνικός έλεγχος θα πρέπει να είναι μια προϋπόθεση, αλλά όχι ο μόνος έλεγχος που θα γίνει, γιατί διαφορετικά η απειλή να παραμείνει η ανάκαμψη μετριοπαθής είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια, κυρία Ορουά, από την Εθνοσυνέλευση της Γαλλικής Δημοκρατίας. και μετά ο κύριος Βίστρομ από την ε, Σουηδία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτό το ε, την ε, συνεδρίαση προβληματισμού για το Ευρωπαϊκό New Deal. Θα πρέπει να υπάρξει εκ νέου εμπιστοσύνη για τις επενδύσεις, όμως καλό θα είναι να αποκτήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και από αυτή την άποψη ο πρόεδρος Σούλτς είπε πριν από λίγο ότι το μόνο οικονομικό κριτήριο δεν, μπορεί, δεν αρκεί και ότι θα πρέπει να προσθεθούν περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες, πράγμα το οποίο βρίσκει σύμφωνα την Εθροσυνέλευση, καθώ σε πρώτη ανάγνωση ενέκρινε νέα κριτήρια, νέου δείκτε πλούτου. Η αύξηση της στόχιας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα πάρα πολύ ανησυχητικό και η κοινωνική διάσταση της οικονομίας θα πρέπει διαρκώς να λαμβάνεται υπόψη. Έχω την εντύπωση ότι από αυτή την πλευρά θα πρέπει να ξεκινήσει ένας συλλογισμός όσον αφορά την, την εισήγηση ενός μήνυμου εισοδήματο σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί χρειάζεται μια εγγύηση πλέον, γιατί το πλάνο Juncker δεν θα φτάσει από μόνο του, δεν είναι το α και το ω που θα λύσει όλα τα προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να έρθω σε αυτό ακριβώ το πλάνο τώρα, τα κριτήρια επιλογής, ακόμα και αν θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που προέβη σε διευκρινήσεις, δεν είναι ωστόσο ακόμα αρκετά σαφή και απλά ώστε να μπορούμε εμείς να είμαστε ήσυχοι όσον αφορά την μόχλευση. Ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων Εντάξει, θα έχουμε και έλεγχο. Ποιο θα είναι ο δημοκρατικό όμω έλεγχο, ο πρόεδρο είπε χτε ότι θα πρέπει πια να φτιαχτεί η ευρωπαϊκή κυβέρνηση και από αυτή την άποψη η δημοκρατική εποπτεία μέσω της εργασίας των κοινοβουλίων θα ενισχυθεί. Όμως δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και θα κλείσω λέγοντας ότι έχω την εντύπωση πως από την άποψη της συγχρηματοδότησης δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά πράγματα που να λένε τι θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα κράτη και ποιες είναι οι διατάξεις που προβλέπονται ώστε να ληφθεί υπόψη ακριβώς οι διορθωτικές πτυχές του Συμφώνου Σταθερότητας. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω με τους ομιλητές εκείνους που επικεντρώθηκαν στην καινοτομία στην Ευρώπη. Γιατί όντως οι καινοτόμοι θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, θα κάνουν επενδύσεις. Πρέπει συνεπώ να είναι ασφαλέστερο και πιο απλό να είναι κάποιος καινοτόμος και επενδυτής στην Ευρώπη μέσα σε αυτούς τους δύσκολους πολιτικά καιρούς που ζούμε. Πράγματι, είναι δύσκολο να δούμε τι μπορεί να είναι πιο απλό, πιο αποτελεσματικό, πιο φτηνό. Και όμως, κυρίως στις, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αναθεωρηθεί το φορολογικό σύστημα. Πολλές φορές οι καινοτόμοι υπερφορολογούνται Πρέπει να έρθουν τα εμπόδια στο επιχειρήν και στις εμπορικές συναλλαγές. Η Ευρώπη δυσκολεύεται, στην Ευρώπη μάλλον πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει κανείς μια νέα επιχείρηση. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε για να έχουμε νέες θέσεις απασχόλησης, αντί να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις παλιές θέσεις απασχόλησης. Είναι βλαβερό σε μια οικονομία να χρησιμοποιούμε επιδοτήσεις για να διατηρήσουμε παλιές θέσεις που δεν έχουν μέλλον. Δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι αυτή η διέξοδος. Πρέπει επίσης να δούμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όλοι λένε ότι χρειάζονται καλύτερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες μέλη και να οθήσουν τις χώρες μέλη προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε όλοι και μετά κυρία Γκίτσοπεκ να ετοιμάζεται. Ο κύριος Όλη παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά από πολλές καθυστερήσεις και παρά τις προς Προσπάθεια του κύριου Γιούνκερ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αποτελέσματα. Περιμένουμε βέβαια επενδύσει από τον ιδιωτικό τομέα. Το επενδυτικό πακέτο το αρχικό είναι βέβαια μικρό σχετικά. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν λοιπόν μέτρα για να διασφαλιστούν κονδύλια για τις οικονομίες των χωρών μελών. Έχω υπόψη μου την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα 60 δισεκατομμύρια το μήνα χρήμα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει όλους τους εταίρους. Επιπλέον θα αποτελέσει ένα κίνητρο για την παραγωγή στην Ευρώπη. Αν επανέλθουμε όμως στο επενδυτικό πακέτο, θέλω να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα. Το βασικό είναι χρήματα στην πραγματική οικονομία. Χρηματοδότηση απευθείας σε βιώσιμα προγράμματα με πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη και για την ε, κοινωνική οικονομία. Δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις για διασφάλιση θέσεων απασχόλησης. Τώρα, όλοι εμείς έχουμε τα εξής ερωτήματα. Πώς θα γίνει η επιλογή, πώς θα τηρηθούν οι βασικές αρχές για να μπορέσει να αναπτυχθεί το δυναμικό και να καταλήξει στην πραγματική οικονομία. Χρειάζονται επενδύσεις στην έρευνα, στην τεχνολογία, σε μικρά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα όμως εδώ να πω ότι θα έπρεπε να γίνουν τα πάντα ώστε να διασφαλίσουμε ότι καμία χώρα μέλος δεν θα μείνει απ' έξω από το πεδίο του επενδυτικού αυτού ταμείου. Πρέπει να υπάρχει καλός συνδυασμός των διαφόρων μέτρων και να απαντηθεί το ερώτημα, διακόπτει ο Πρόεδρος, ολοκληρώνω. Υπάρχει καμία εκτίμηση για το αποτέλεσμα όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και θα έπρεπε η απάντηση να δείξει τελικά τι θα πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και αν αξίζει τον κόπο η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ε, ε, Από τη Σλοβενία παρακαλώ. Και να ετοιμάζεται το επόμενο ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Σλοβενία έχει αναπτύξει δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι ευρωπαϊκοί πόροι. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει το δρόμο για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημοσιονομική ε, προσαρμογή και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να υποστηρίξουμε ως Σλοβενία το επενδυτικό σχέδιο. Ιδιαίτερα στην κατεύθυνση που ήδη κατεγράφει. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική με τα μέτρα και τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις είναι η σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα είναι να συνενωθούν όλα αυτά τα μέτρα και να κατευθυνθούν προς τον ίδιο κοινό στόχο. Μια από τις θετικές πτυχές αυτού του σχεδίου είναι ότι δεν αφορά μόνο οικονομικά μέτρα ή μέσα, αλλά και τεχνικά μέτρα, μέτρα τεχνογνωσίας, κέντρα παροχή συμβουλών. Βέβαια, δυστυχώς ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα η δομή τους, η λειτουργία τους και η χρηματοδότησή τους. Γιατί υπάρχει μια σειρά από ε, δομές ήδη και δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η ίδια δουλειά. Εάν θέλουμε λοιπόν ένα νέο ε, κέντρο παροχή συμβουλών πρέπει να επιτρέψουμε τη συμμετοχή σε αυτό όλων των εθνικών επενδυτικών τραπεζών και να συνενώσουμε όλη την καλή δουλειά που ήδη γίνεται στο τομέα αυτό. Κριτήρια για την έγκριση των σχεδίων πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν θα επιβάλλει διακρίσεις εις βάρος των μικρότερων ή πιο αδύναμων κρατών μελών. Ούτε και θα πρέπει να βρίσκονται σε δημισμενέστερη θέση ε, κράτη ε, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν γίνει οι κατάλληλε επενδύσεις στις υποδομές ακόμη. Αντιθέτω, πρέπει αυτά τα μέτρα να είναι συμπληρωματικά ως προσυφιστάμενα μέτρα και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω πως η εθνική συνεισφορά μαζί με, τον, με την αντιμετώπιση του εθνικού ε, ελλείμματος θα πρέπει να προχωράει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ την συνάδελφο από τη Λιθουανία. Τον συνάδελφο από τη Λιθουανία και να ετοιμάζεται η κυρία Κέλογαν. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θυμόμαστε από την από τα μαθητικά θρανία μας και το μάθημα της φυσικής. Το όνομα της αδράνειας, ότι δεν αλλάζει η ενέργεια, δεν εξαφανίζεται η ενέργεια, μόνο αλλάζει η μορφή. Ε, το ίδιο μπορούμε να το διαπιστώσουμε και στην οικονομία. Το χρήμα δεν, δεν χάνεται, απλώς αλλάζει τσέπη. Εχθές αναφέρθηκε ότι το 1% των πιο πλούσιων του κόσμου έχουν ενισχύσει έχουν αυξήσει την περιουσία τους κατά τρόπο πολύ, πολύ ε, ουσιαστικό. Το επενδυτικό σχέδιο λοιπόν του Juncker προσφέρει τη δυνατότητα 5 δις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 16 δις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με συνολικό όγκο 300 δις επενδύσεων. Πολύ ωραία το υποστηρίζουμε, ιδιαίτερα εάν πρόκειται να ενισχυθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στόχοι όμως πρέπει να είναι οι εξή. Στόχοι θα είναι να μην χάσει τον προσανατολισμό του ευρωπαϊκός προπολογισμό του βασικού στόχου της στρατηγικής του 2020, τον ορίζοντα, το πρόγραμμα για τον ορίζοντα, το κοινωνικό τομείο δεν θα πρέπει να λησμονούμε τις στοχευμένες εκείνες δαπάνες που θα φέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα γιατί θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά τα περιμένει όχι μόνο το 1% των πλουσίων αλλά και το υπόλοιπο 99% των μη πλουσίων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε πώς θα διανύμουμε, πώς σε, αυτό θα πρέπει να βρούμε πώς θα διανύμουμε τους σπόρους. Σας ευχαριστώ. Κέλλερ. Και μετά Σαφοζέχ για να δώσουν στη συνέχεια τις απαντήσεις οι ομιλητές μας και να ξαναγυρίσουμε σε ερώτα απαντήσεις. Κέλλερ. Ονομάζομαι Κέλλερ. Είμαι από την Γερουσία στο Παρίσι. Αλλά είμαι από το Στρασβούργο. Και είμαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στο ε, ημικύκλιο των Βρυξελών, ενώ το η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι στη πόλη μου, το Στρασβούργο. Όλοι διαβάσαμε το σχέδιο Juncker που στόχο έχει να αναζωπηρώσει τις δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις και πολλοί συνάδελφοι είπαν πόσο λογικό είναι αυτό ε, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα ήθελα κυρίω να προσθέσω για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και μιας νέα ελπίδα για τους ε, Ευρωπαίους νέους. Όμως μένουν σημεία που πρέπει να να διευκρινιστούν. Η ε, ισχύς του της μόχλευσης που αναμένεται θα πρέπει να δούμε πόσο θα υλοποιηθεί. Αυτός ο πολλαπλασιαστής του 2015 θα πρέπει να τεκμηριωθεί και αν μου επιτρέπετε κύριε πρόσωπε της ΕΤΕΠ δεν είναι ακριβώς το ίδιο το να δίνουμε ίδιου πόρους σε μια τράπεζα με προφανές εφέ μόχλευσης στον όγκο πιστώσεων που χορηγεί και να κάνουμε διάφορα μοντάζ με αυτόν τον συντελεστή πολλαπλασιαστή Δεύτερον, τα κρατη που δεν ξέρουμε πώς θα χρηματοδοτηθούν, τα κράτη-μέλη που αποκλείονται που μάλλον που οι επενδύσει των κρατών μελών που αποκλείονται από τον υπολογισμό. Ε, Πώ ακριβώ θα γίνει αυτό στην πράξη. Τρίτη ερώτηση. Τι γίνεται με εκείνα τα προγράμματα που μπορεί να είναι κοινοτόμα, αλλά με χαμηλότερο εφέ μόχλευση, για παράδειγμα, στο τομέα τη έρευνα. Ας πούμε, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα θεωρούνται τομείς ε, καινοτόμοι και με δυναμικό. Και τέταρτη μου ερώτηση, ποιοι θα είναι οι τρόποι επιλογής των προγραμμάτων, ποιος θα είναι ο ρόλος των κρατών μελών, ποιος θα είναι ο ρόλος ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Στρατικές Επενδύσεις, ποια θα είναι η διακυβέρνησή του και Καθώς η συνάδελφος, μάλλον όπως και η συνάδελφος Φερέιρα, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η ανάλυση κινδύνου, κυρίως στις ε, χώρες που έχουν ευαισθητοποιηθεί λόγω της ε, κρίσης. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, αλλά και ο, το εφέ μόχλευσης μεγαλύτερο. Ευχαριστώ. Σαφχάουζερεν τώρα. Δεύτερο Στρασβούργο, Γέζος. Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώ, φοβόμαι πως αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων και ανάπτυξη δεν θα λειτουργήσει. Ε, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αν είχαμε θελήσει να βγούμε από την ύφεση και από την κρίση του ευρώ, θα χρειαζόταν να επενδύσουμε κατά προτεραιότητα στις χώρες που διαρθωτικά είναι ελληματικέ. Και το θέμα των επενδύσεων προ τέτοιε χώρες είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί διαφορετικά θα αποκατασταθούν οι λογαριασμοί μας μέσω της ύφεσης, της ανεργίας αλλά και της κοινωνικής κρίσης και τέλος της διάλυσης της Ευρωζώνης. Αλλά για να γίνουν επενδύσεις στις διαφορετικά ελληματικές χώρες θα χρειάζονταν προγράμματα τα οποία θέλουν προετοιμασία, δεν ε, ε, γίνονται από μόνα τους, πρέπει να οικοδομηθούν πιο συγκεκριμένα με βάση την πράσινη οικονομία και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχουμε ποσά τα οποία θα αντιστοιχούν όχι σε κεφάλαιο και σε, και μόχλευση αλλά σε πραγματικά μέσα που θα αντιστοιχούν σε αυτό που θα ήταν ένα, μια χαλάρωση, μια ποσοτική χαλάρωση, όχι για να σωθούν τράπεζες και να αγοραστούν ε, χρέη, δηλαδή να φτιάξουμε χρήμα, αλλά για να επενδύσουμε σε προγράμματα πραγματικά αποδοτικά. Αυτή τη διάσταση την οποία εμείς θα θέλαμε να, να προχωρήσουμε με τον Μάντι, τον Βασανίνη και αυτή τη διάσταση λοιπόν τελείωσε, την, την εγκαταλείψατε και αυτό είναι πραγματικά κρίμα και ζημιογόνο γιατί δεν θα καταλαβαίνω πώς θα δημιουργήσετε αυτό το φεμόχλευσης αν δεν επενδύσετε μαζικά στις διαρθωτικά ελληματικές χώρες και δημιουργώντας ή μάλλον προετοιμάζοντας προγράμματα και επιτρέποντας την πράσινη οικονομία να αναπτυχθεί. Το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα της εμπιστοσύνης, ούτε το πρόβλημα της νομοθεσίας. Το πρόβλημα είναι οι επενδύσεις στις ελληματικές χώρες. Δεν απαντάτε σε αυτό και η αγορά δεν θα σας ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το πάνελ μας τώρα. Ο κύριος Μόρτερ πρώτα, επειδή πρέπει να φύγει σε λίγο και μετά ο Επίτροπος Μοσκοβισή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για το μέγεθος. Θα σας δώσω μια έδειξη. Φυσικά και μαζί με την Επιτροπή ρωτήσαμε τα κράτη-μέλη για τις δυνατότητες. Και υπάρχει αυτός ο περίφημος κατάλογος που μιλάει για 1,3 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Εμείς βέβαια το κοιτάμε, οι εμπειρογνώμονες. Είναι ποσά που πρόκειται να επενδυθούμε μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Που θα καταλήξουν στα 500 δισεκατομμύρια. Τα 315 δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά. Δεύτερον, είναι μέρος των επενδύσεων, γιατί η ΕΤΕ, όπως κάνει πάντα, θα συνεχίσει. Μιλάμε για επιπλέον όγκο επενδύσεων αυτών του πακέτου Juncker. Έτσι κι οι δημόσιες επενδύσεις είναι πάντα ε, το, ο κύριος παράγοντας των συνηθισμένων μας επενδύσεων. Πρέπει να αρχίσουμε λοιπόν με αυτό και να δούμε ποια θα είναι η εμπειρία μας. Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε μια διάκριση ανάμεσα στο ποιοι είναι οι τομείς που επιλέγονται, που είναι οι μεταφορές, οι υποδομές, η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές, τα κοινωνικά υποδομές κλπ. Να κάνετε διάκριση ανάμεσα στους τομείς λοιπόν και τα προγράμματα που επιλέγονται. Γιατί οι τομείς είναι κάτι διαφορετικό από την επιλογή των προγραμμάτων αυτών καθεαυτών. Οι ιδιωτικοί επενδυτές θα συμμετάσχουν όταν θα έχουν γίνει σοβαρά και καλά αυτά τα πράγματα από επαγγελματίες και βέβαια αυτή τη δυνατότητα την προσφέρουμε εμείς από την ΕΤΕ. Γιατί τα προγράμματα πρέπει να είναι υγιή τραπεζικά μιλώντας και τεχνικά και οικονομικά δηλαδή και τεχνικά. Για μένα λοιπόν η διάκριση αυτή έχει τεράστια σημασία. Στη συνέχεια έχουμε τους τρεις πυλώνες. Και να το λάβετε αυτό υπόψη σας. Πρώτον, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό καλύπτει και από τη startup και από κεφαλακές και μικροχρηματοδοτήσεις μέχρι τη χρηματοδότηση της ε, καινοτομίας και μεγάλους συνετορισμούς. Φυσικά υπάρχει και το δεύτερο σκέλος που είναι η καινοτομία αυτή καθεαυτή. Εκεί μπορούμε να αναλάβουμε υψηλότερους κινδύνους μια που υπάρχουν οι πρώτες εγγύσεις και άρα εδώ μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις για την καινοτομία. Και οι υποδομές είναι και οι πληροφορικοί και οι γενικότερες υποδομές. Και το τρίτο είναι το εξή. Έχουμε συμπεριλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Jaspers και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε το πεδίο και τις δυνατότητες. Γιατί σίγουρα οι ανάγκες είναι τεράστιες σε πολλές χώρες μέλη. Για τον πολλαπλασιαστή τώρα. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι μάλλον συντηρητική και βασίζεται στην μέχρι τώρα εμπειρία μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε αυτό λεπτομερώς. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και θέλω να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Πρώτον, από την νομοθεσία αυτή καθεαυτή γιατί η ποιότητα των εγγύσεων είναι στοιχείο κλειδί για τις επενδύσεις και θα εξαρτηθεί βέβαια και από την ποιότητα των προγραμμάτων γιατί ανάλογα με το πόσο καλά είναι θα προσελκύσετε περισσότερες ή λιγότερες επενδύσεις. Αυτά είναι στοιχεία κλειδί για τον πολλαπλασιαστή. Το περιφερειακό τώρα σκέλος θέλω να τονίσω και αυτό. Ποιες είναι οι πέντε κύριες χώρες των δραστηριοτήτων μας. Είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία. Βλέπετε ότι είναι από τις χώρες που αναφέρατε. Δραστηριοποιούμεθα λοιπόν και στις χώρες προγράμματος. Αυτό τώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι να έχουμε τη συνολική εικόνα. Εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας γενικότερης στρατηγικής. Η πρωτοβουλία για την κεφαλιακή αγορά αποτελεί μέρος μιας τέτοιας, ενός τέτοιου συνολικού σχεδίου. Εφόσον προσελκύουμε κεφάλαια στην Ευρώπη, ενισχύουμε και το πακέτο Juncker. Μαζί πρέπει να τα δούμε αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως σας είπα, η τράπεζά μας είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει. Χρειαζόμαστε υγιή, σαφή ε, νομοθεσία, αριθμιστικό πλαίσιο για την πρωτοβουλία Γιούγκερ και χρειαζόμαστε επαγγελματίες συνομιλητές και από πλευράς του δημοσίου και από πλευράς του ιδιωτικού τομέα με καλά σχεδιασμένα και καλά εφαρμοσμένα προγράμματα. Αυτά χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μορτέ. Τώρα ο Επίτροπος Μοσχοβησί έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ο Πρόεδρος, ο ε, της ΕΤΕΠ απάντησε στο το των ερωτήσεων που μας υποβλήθησαν η πρώτη ερώτηση ήταν ε, κατά πόσο θεωρούμε πως είναι ανεπαρκές αυτό το πλάνο επενδύσεων. Αυτό το, το ακούω από όλες τις πλευρές ε, όσον αφορά τις αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν ε, όσον αφορά το σχέδιο Juncker. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ορίζοντας το σχέδιο επενδύσεων μαζί με την ΕΤΕΠΕ λάβαμε υπόψη την τρέχουσα κατάσταση των δημοσίων οικονομικών, της δημόσιας οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη έχω την πεποίθηση και αυτό μπορούμε να σας το αποδείξουμε με τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει πως πρόκειται για ρεαλιστικό ε, σχέδιο και να σας πω ταυτόχρονα ε, τα εξή. Πρώτον, πιστεύω πως είναι αλήθεια ότι το Ταμείο θέλουμε να έχει σημαντική μόχλευση, αλλά έχουμε φτάσει και το μηχανισμό διακυβέρνησης που θα μας επιτρέψει να το επιτύχουμε αυτή τη μόχλευση και ότι ό,τι φαίνεται στο πλαίσιο της ΕΚΤ ε, είναι πολλά υποσχόμενη κατάσταση. Φυσικά θα πρέπει να το παρακολουθούμε αυτό και εσείς εδώ από το Ευρωκοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είμαι βέβαιος ότι οι ανάγκες επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 315, 300 ε, 75 δις. Αλλά, μη, αλλά φανταστείτε ότι πρόκειται για σύντομη διαδικασία. Έξι μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να λειτουργούμε. Δηλαδή, στην ουσία σε δύο χρόνια θα διαπανίσουμε 300 τόσα εκατομμύρια. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το ποσό και αν όντως αποδειχθεί επιτυχές και το είπε και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εδώ ότι θα είναι επιτυχές τότε θα μπορέσουμε να παρατείνουμε αυτό το πρόγραμμα. Στην πράξη θα έχουμε 100 δις επιπλέον για καμιά δεκαετία. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Είναι το πρώτο στάδιο αυτό. Δεύτερον, για την επιλογή των σχεδίων και τα όσα είπατε. Η διαδικασία θα είναι διαφανής, θα εξασφαλιστεί από ένα είδος ε, ε, task force και αυτό που το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα πρόκειται όντω για επιπλέον επενδύσει και στοχοθετημένε επενδύσει στου τομεί που διευκρινίσαμε. Και εδώ και πάλι με, διευκρινί... με... με περισσότερε λεπτομέρειε ε, ε, στη συνέχεια. Βεβαίω συνειδητοποιώ τι παρατηρήσει που κάνατε ε, για το γεγονό ότι θα πρέπει ταυτόχρονα, χωρί να υπάρξει ε, ε, δίκαιη επιστροφή, να λάβουμε υπόψη τι χώρε που έχουν μεγαλύτερε δυσκολίε. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο, η ευελιξία όπως την ορίζει η Κομισιόν εφαρμόζεται για τις, τις χώρες που βρίσκονται στο προληπτικό σκέλος παρά στο διορθωτικό και εδώ δεν νομίζω πως είναι παράλογο αυτό γιατί αν είχαμε φτιάξει ένα σχέδιο που θα απομάκρυνε από το σύμφωνο σταθερότητας όλες τις επενδύσεις όπου και αν αυτές γίνονταν τότε δεν θα υπήρχε πλέον ε, σύμφωνο δεν θα υπήρχε καμία παρότρινση στις μεταρρυθμίσεις, για μεταρρυθμίσεις ενώ εμείς θέλουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση Αλλά βέβαια θα πρέπει να είστε βέβαιοι πως βεβαίω θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες εξυγχρονισμού των οικονομιών που διατρέχουν κρίση μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων και εκεί θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να, γεννηθούν και να αναπτυχθούν βιώσιμα προγράμματα. Θα ήταν τρελό τα, τα κονδύλια να πάνε πρώτα σε χώρε οι οποίε είναι σε καλή κατάσταση αντί να πάνε στι χώρε ε, που ε, υποφέρουν περισσότερο ή ακόμα και αν δεν είναι πολιτικοί, αυτοί οι, οι που θα τα αποφασίσουν και θα τα εγκρίνουν θα, θα το έχουν αυτό υπόψη τους. Το σχέδιο αυτό θέλουμε να κινητοποιήσει ε, την ανάπτυξη αλλά και τις επενδύσεις. Ξέρω πως έχουν γίνει ήδη αξιολογήσεις, οι οποίες ε, είναι μάλλον αισιόδοξε. Εγώ εξακολουθώ να τις εξετάζω με ε, μεγάλη σύνεση, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε κάνει διαρκώς αξιολογήσεις, γιατί Τελικά περί αυτού πρόκειται. Ε, έλλειμμα επενδύσεων, έλλειμμα ανάπτυξης, έλλειμμα απασχόλησης. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με μια Ευρώπη που διαρκώς είναι στο 1% της ανάπτυξης, στο 1% του πληθωρισμού. Και εδώ χαιρετίζω και ένα επιπλέον ε, τομέα που είναι η δράση της ΕΤΕΠ και με ε, τεράστιες ανισότητες και τεράστια ποσοστά ανεργίας. Αν συνεχίσει να λειτουργεί έτσι η Ευρώπη δεν θα υπάρχει μέλλον. Και ακριβώς το να φτιάξουμε ένα σχέδιο επενδύσεων, τι είναι οι επενδύσεις ένα στοίχημα στο, για το μέλλον. Ένα στοίχημα το οποίο θέλουμε να ε, περιχαρακώσουμε με στέρεους και συμπαγείς μηχανισμούς και μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρτουή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρισκόμαστε ενώπιον της μελέτης του σχεδίου νομοθετήματος που θα ορίσει νομική βάση για την υλοποίηση του σχεδίου Juncker. Άρα η σημερινή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχει τεράστια σημασία για να λάβουμε υπόψη τις δικές σας ε, παρατηρήσεις, ε, τα ερωτηματικά, τους προβληματισμούς σας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα τα λάβουμε υπόψη όλα. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι εδώ έχουμε εγγυήσει πάνω σε αυτέ τι το σχέδιο, εγγυήσει οι οποίε θα πρέπει να εγκρίνει με την ψήφο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγγυήσει οι οποίε απαιτούν την εισφορά πόρων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, πιστώσεων τις οποίες θα πρέπει να αντλήσουμε από προγράμματα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 και όπου πάρουμε 10 θα δώσουμε πίσω το δεκαπλάσιο, 150, χάρη στη μόχλευση. Αυτό πρέπει να επαληθευτεί φυσικά. Έχω κάθε ελπίδα ότι η εγγύηση θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις όπως τη χρειαζόμαστε. Η εγγύηση αυτή προϋποθέτει ότι θα είναι διαθέσιμη η πόρη... Και μια και εκπροσωπείται Εθνικά Κοινοβούλια, θα ήθελα να σας επισημάνω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει να σωρεύονται εδώ και χρόνια ανεξόφλητοι λογαριασμοί και πρέπει τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να είναι τόσο επιφυλακτικά ως προς τη διάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πιστώσεων που χρειάζονται για να εξοφληθούν εκρεμείς λογαριασμοί. Λέγοντας αυτό και απαντώ στην κυρία Κελέρ για την έρευνα, ότι ρε ναι, βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή εδώ γιατί υπάρχουν ερευνητικά κέντρα τα οποία δεν είναι σε θέση να ε, καταφύγουν στον δανεισμό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ούτως υπήν, ούτως, άρα θα πρέπει να κάνουμε ε, μία ρύθμιση αρκετά προσεκτική που να κάνει τη διάκριση και να επιτρέπει τη χρηματοδότηση. Εγώ είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω πέρσι με τον πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το προσέξουμε ιδιαίτερα. Βεβαίως η εδαφική πτυχή θα έχει μεγάλη σημασία. Το Ταμείο ε, Συνοχής σημαίνει ότι περιοχές που έχουν ανάγκη από συγκεκριμένε υποδομέ μπορούν να αντλήσουν τους πόρους που διαθέτει το σχέδιο Juncker προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους ώστε η ανάπτυξη και η απασχόληση να ε, υλοποιηθούν όπως το προσμένουν. Ο πρόεδρος Ρεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρτουά. Έχουμε τον κύριο Ντόνελεν, τον κύριο Ντόνελη πρώτο και μετά τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβούλιο. Κύριο Ντόνελη, πρόεδρε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα και αλλά και στη χθεσινή συνεδρία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη και την απασχόληση με το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων και την ποσοτική χαλάρωση ως μέσα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διαθέσει πολύ φθηνό χρήμα στους ε, επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα στηρίξει τον κίνδυνο, θα καλύψει τον κίνδυνο των επενδύσεων. Αυτό προβλέπει ως εκ τούτου μια αύξηση του ΑΕΠ μέσω πρόθεσμα και ε, ανάπτυξη του αριθμού των θέσεων εργασία. Ελπίζουμε αυτή η ποσοτική χαράλωση να μην οδηγήσει σε φούσκα και να μην επιβαρύνει τη θέση των πιο φτωχών. Οι επενδύσεις της ΕΤΕΠ στηρίζονται στις, στο κέρδος, που σημαίνει κέρδος και απόδοση στις μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή στους κεφαλαιούχους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με σχέδια που θα πρέπει να υποστηριχθούν, που δεν είναι απαραίτητα βιώσιμα εμπορικά. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ε, κέρδος από επενδυτικά σχέδια όπου αναλαμβάνει τον κίνδυνο ο πολίτης γιατί ο ιδιωτικό τομέα δεν τα κρίνει οικονομικά ή εμπορικά βιώσιμα. Ερωτώ λοιπόν, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δύο αυτά μέσα προκειμένου να ενισχύσουμε τις θέσεις εργασίας μέσο και μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουμε θέσει εργασία, να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι το οικονομικό όφελο από τα δύο αυτά μέσα θα το ε, εισπράξουν όχι μόνο οι πιο ε, εύρωστοι οικονομικά, όχι μόνο οι πιο πλούσιοι, αλλά όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι οι πολίτε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να φροντίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την εισαγωγή παραδείγματι ενό φόρου επί, της επί του ωφέλου αυτών των δύο δραστηριοτήτων τη ΕΤΕΠ και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή το κέρδο που θα παράγεται θα πρέπει να φορολογείται στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να χρηματοδοτεί το ε, δημόσιο κέρδος και άρα μπορούν τα χρήματα αυτά στη συνέχεια να χρηματοδοτούν δημόσιες επενδύσεις όπως ευρυζωνικότητα, εκπαίδευση, υποδομές κτλ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, δεν μπορώ να σας περισσότερο χρόνο. Ο κ. Ζιούκ από το Βέλγιο και μετά ο κ. Βέστλουντ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θετικά βλέπουμε εμείς το επενδυτικό αυτό σχέδιο, παρόλο βέβαια που αναρωτιόμαστε γιατί δεν χώρες μέλη να επενδύσουν στα πλαίσια του πακέτου ανεξιοδιών. Ε, αναρωτιέμαι για τα ποσά, για τη μόχλευση, για την υποκατάσταση άλλων προγραμμάτων. Η κύρια όμως ερώτησή μου έχει να κάνει με τον ίδιο τον προσανατολισμό του επενδυτικού αυτού σχεδίου. Ο κύριος Μοσχοβησή ήταν κάπως πιο συγκεκριμένος για τους στόχους του και πολλά από αυτά μου ακούγονται θετικά, ανανόσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση. Όμως διατηρώ την εντύπωση ότι έχουμε βάλει λίγο απ' όλα στους στόχους μας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η απασχόληση φυσικά και είναι κεντρικό ζήτημα. Από την αρχή πρέπει να είναι κριτήριο και όχι στην αξιολόγηση. Να είναι δηλαδή κριτήριο τα προγράμματα που συζητάμε για να επιλέξουμε δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει και για το περιβάλλον. Εν μάλιστα και της διάσκεψης του Παρισιού. Η ενέργεια που είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Ελπίζω λοιπόν όσο συνεχίζονται οι εργασίες ο στόχος να γίνει πιο συγκεκριμένος. Τέλο για το New Deal, τη νέα συμφωνία, γιατί πολλοί μα λένε ότι το πακέτο αυτό το επενδυτικό Juncker είναι το New Deal τη Ευρώπη. Σε εκείνο του Ρούσβελτ δεν υπήρχαν μόνο επενδύσει. υπήρχε και οικονομική ρύθμιση. Ε, διακρίναμε τι τραπεζικέ δραστηριότητε από την κοινωνική συνοχή. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε επενδυτικό πακέτο αν δεν υπάρξει τέτοια δημοσιονομική ρύθμιση, αν δεν αλλάξει το τραπεζικό σύστημα ώστε να επενδύουν στην πραγματική οικονομία και αν δεν προσέξουμε όλος ιδιαίτερος την κοινωνική διάσταση. Αν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ε, του καταναλωτή ούτε του επενδυτή και άρα δεν θα λειτουργήσει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βέστλουντ είναι ο επόμενος και ο κύριος Μπελετζεύσκη από την Πολωνία. Να ετοιμάζετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το επενδυτικό αυτό σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Στην Riksdag, στη Σουηδία, το έχουμε συζητήσει και έχουμε καταλήξει πολύ συγκεκριμένα. Είμαστε θετικοί, προσεκτικοί συγχρόνως. Δεν έχουμε απάντηση σε όλα, καθ' άλλο. Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων είναι κάτι που ακόμα συζητάμε. Έχω την αίσθηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα για το τι προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν. Ακούω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που λέει ότι θέλει να συζητήσουμε τα προγράμματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως δεν είναι αυτό που δίνει χρήματα, ελέγχει τον προπολογισμό, αλλά όχι τα προγράμματα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι θα γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι θα έπρεπε να ακούει τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα έχουν λόγο. Και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έπρεπε να ακούνε τα εθνικά κοινοβούλια. Να ξέρουν τι συζητάνε. Θα ήταν σημαντικό βρίσκω. Γιατί έτσι θα γινόταν κατανοητό ότι δεν πρόκειται για ένα ομόσπονδο κράτος η Ευρώπη, αλλά ένα φόρουμ συνεργασίας μεταξύ 28 χωρών μελών που πρέπει να μπορούν να έχουν λόγο και ο λόγος τους αυτός να γίνεται σεβαστός. Ο κύριος Γαλαζένσκι, Πολωνία, είναι επόμενος ομιλητής και μετά ο κύριος Γιούγκ, την Αλληλική Εθνοσυνέλευση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε μια ιδέα που ακούστηκε ήδη και προτάθηκε από τον κύριο Αρτουή, αν δεν απατώμε. Πρόκειται για μια διάκριση που πρέπει να γίνει ανάμεσα στις χώρες που έχουν το ευρώ και σε εκείνες που δεν έχουν το ευρώ. Οι χώρες που έχουν το ενίο νόμισμα θα μπορούσαν να έχουν μια περίπου κυβέρνηση. Έχουμε βέβαια, εγώ θα σας θυμίσω, μια κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ρωτώ, πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Πρόεδρε, μια άλλη επιτροπή σκέφτεσαι, μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ασχολείται μόνο με την Ευρωζώνη και τότε αυτή η παλιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουμε τώρα που ασχολείται με όλες τις χώρες μέλη, τι θα έκανε. Και αν ε, συνεχίσουμε στην λογική αυτή, τότε θα πρέπει να έχουμε και ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να ασχολείται μόνο με τις χώρες της Ευρωζώνης. Εκτός ευρώ υπάρχουν οικονομίες που είναι σημαντικές, όπως η Φιλανδία. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα ήταν ε, καλή ιδέα. Εμείς πάντως είμαστε κατά και πιστεύουμε ότι έτσι καταλήγουμε και σε κάτι άλλο. Αν θέλουμε να διχάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξέρετε ότι αυτό ακριβώς θέλουν όλα τα λαϊκά, ε, όλα τα λαϊκίστικα κινήματα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Επόμενος, ο κύριος Γιούγκ και μετά να, κοιμάζ, ετοιμάζεται από την Πορτογαλία ο κύριος Σαφτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για το πρώτο σκέλος της συζήτησης πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον. Σήμερα συζητήσαμε πολύ για το πακέτο Juncker. Βέβαια υπάρχει και κάτι παράδοξο εδώ. Γιατί τα προγράμματα λιτότητας που εφαρμόσαμε εμεί στη Γαλλία για παράδειγμα είχαν σαν αποτέλεσμα να επιβραδύνουν τις επενδύσεις, τις δημόσιες επενδύσεις και πάρα πολύ τις επενδύσεις των τοπικών αρχών. Οπότε χαίρομαι που τώρα αλλάζουμε δρόμο. Μία από τις ερωτήσεις μου όμως είναι η εξής. Λέτε ότι θέλετε συνεισφορές από τις χώρες μέλη σε αυτό το ταμείο, το επενδυτικό με τα 315 δισεκατομμύρια. Ωραία, είναι καλή ιδέα. Όμως, σκέφτομαι το εξή. Πού θα τα βρούμε εμείς αυτά τα χρήματα. Δεν θα τα δανειστούμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ήταν πολύ παράδοξο αυτό. Συνεπώς ρωτάω, τι έχετε στο μυαλό σας. Εντάξει, οι χώρες θα σας απαντήσουν, αλλά εσείς με την πρότασή σας τι υποθέτετε, πώς νομίζετε ότι θα ανταποκριθούν οι χώρες, με τι μέσα. Έχετε καμιά ιδέα για τα ποσά τα οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει κάθε χώρα. Για το δεύτερο τώρα τμήμα της συζήτησης πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι σε ένα μεγάλο βαθμό τις απόψεις του Πρόεδρου της Επιτροπής Προπολογισμών, του κυρίου Αρτουή, για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, για την ανάγκη να έχουμε μια ισχυρή διακυβέρνηση με έναν Υπουργό Πλήρους Απασχόλησης και μια διεύθυνση και ένα ταμεία που να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως όλα αυτά είναι στην σφαίρα των υποθέσεων, είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Και μια από εδώ βρισκόμαστε στα πλαίσια του άρθρου 13, τουλάχιστον έτσι λέει η μερίσια διάταξη, Ερωτώ, πώς θα προχωρήσουμε για να θέσουμε σε εφαρμογή το άρθρο 13. Χτες ακούσαμε μόνο τις προτάσεις του κύριου Σαραζάν από την Γερμανία που έκανε τρεις-τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του άρθρου 13. Μα νομίζω ότι αυτό πρέπει να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις επ' αυτού και να βγούμε από αυτή την αίθουσα έχοντας στο νου μας διάφορες ιδέες και προβληματισμό. Ευχαριστούμε κύριε Γιόγκ. Επόμενος, ο κύριος Σάφρα από την Πορτογαλία. Η κυρία Καπριέλ Κρετού από τη Ρουμανία θα είναι η ομιλήτρια μετά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου, τα χαμηλά επίπεδα, επίπεδα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων δεν επιτρέπουν σημαντική και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Αλλά δεν ε, ωφελεί να μιλάμε για επενδύσει, μιλά... αλλά πρέπει να δημιουργηθούν οι προποθέσει ώστε να γίνουν οι επενδύσει. Στην Πορτογαλία η εφαρμογή τη πολιτική λιτότητα που επιβλήθη από την ε, τρόικα ε, οδήγησε τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις στα χαμηλότερα πεδία από ε, εδώ και 25 χρόνια. Ε, θα ξεπεραστεί δε το χρέος, ε, το χρέος αυξάνεται ε, ενώ αντιστρόφως ανάλογα μειώνονται οι επενδύσεις. Ε, η δημοσιονομική εξυγένση οδήγησε σε μετατροπή της ιστορικής ζήτησης ε, και άρα την μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Με την λιτότητα και με την δημοσιονομική εξυγίαση, οι ιδιωτικέ και οι δημόσιε επενδύσει έχει φτάσει στην Πορτογαλία στα χαμηλότερα επίπεδα στην πρόσφατη μα ιστορία. Μετά από βαθιά ύφεση, η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή είναι ανεμική και δεν υπάρχουν προοπτικέ να βελτιωθεί. Πέρα από το πρόγραμμα της ε, Τρόικα, παρότι το εφαρμόσαμε, η, η Πορτογαλική κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει τη λιτότητα ε, και με βάση αυτό ε, το σύμφωνο, το δημοσιονομικό, το οποίο υποτίθεται είναι εγγύηση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Όμως ε, τα μέτρα αυτά δεν είναι βιώσιμα και ακόμα και μια απόπειρα επιτευξή θα οδηγούσε στην τελμάτωση την οικονομική και σε επίπεδα ακόμη ψηλότερη ανεργίας. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, πιστεύουμε ότι αυτό το σύμφωνο θα πρέπει να προβλέψει συγκεκριμένα προγράμματα στήριξης για τις χώρες οι οποίες έχουν μπει σε προγράμματα για να μπορέσει να παγιωθεί μια οικονομική ε, πολιτική για να προωθηθεί η ανάπτυξη αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις χώρες αυτές. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Κρέτσου. Και μετά η κυρία Χέλμαν επένω να ετοιμάζεται παρακαλώ. κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί φίλοι. οργανωτή και οι κύριοι ομιλητέ σήμερα μα γέμισαν μαύρο χιούμορ και αναπάντεχη ειλικρίνεια. Μας επαναλαμβάνουν δηλαδή διαρκώς με φωνή γεμάτη κύρος ότι ζούμε σε μια οικονομία, σε μια αγορά. Εμείς είμαστε βουλευτές εδώ και εκπροσωπούμε τον Ευρωπαίο πολίτη. Παλαιομοδίτικο πολίτη που εξακολουθεί να πιστεύει ότι ζει σε μια κοινωνία όπου η στέγη, η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία βοηθούν τον άνθρωπο και την κοινωνία του. Και είναι τα θέματα πάνω στα οποία πρέπει να συζητούμε και να λαμβάνουμε αποφάσεις. Η κοινωνία της αγοράς, είναι ήδη αρκετά τρομακτική για τον πολίτη. Τους φαίνεται αδιανόητο να τους λέμε μόνο ότι ζουν σε οικονομία αγοράς. Δεν τους βοηθάμε λοιπόν να, την, ε, να το κατανοήσουν αυτό. Αυτό το διαπιστώνουμε και πολύ ημών. Διαπιστώνουμε μαύρο χιούμορ όταν μιλάτε για ευρωπαϊκό ιδεώδες. Αγαπητοί φίλοι, όταν ξεκίνησε με το ιστορικό εκείνο πρόγραμμα ο Ρούσβελτ, ο Ρούσφελτ είπε σε ολόκληρο το έθνος, άνδρες και γυναίκες λησμονημένοι από την πολιτική φιλοσοφία του συστήματος, στρέφουν σε μας το βλέμμα για περισσότερες και πιο ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής στην κατανομή του εθνικού πλούτου. Δεσμεύομαι λοιπόν σε ένα New Deal, σε μια νέα συμφωνία για τον Αμερικανικό λαό. Πέρα στις παραθέσεις. Αγαπητοί φίλοι, ο Μάρξ έγραψε κάποτε η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία, τη δεύτερη ως φάρσα. Και φοβούμε ότι είχε δίκιο. Ξεχάσαμε να πούμε τη φράση «Δεσμευόμαστε σε ένα νέο deal για τις ευρωπαϊκές αγορές». Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής, επόμενη ομιλητρία, η κυρία Χέλμα Νέπενος και παρακαλώ τον κύριο Χέλμουτ Μαρκού να ετοιμάζεται. Πρόεδρε, είμαστε θετικοί με την ιδέα αυτή του επενδυτικού ταμείου, αλλά είμαστε επικριτικοί στην Ολλανδία γιατί έχουμε διάφορες ερωτήσεις. Τι θα κοιτάξουμε, τα στάνταρ προγράμματα δεν θα έπρεπε να κοιτάξουμε περισσότερο τα καινοτόμα, αυτά που έχουν να φέρουν κάτι καινούριο στην οικονομία. Αυτό είναι ζωτική ε, ε, σημασία για μα. Και αν το κάνουμε, μιλάμε για 315 δισεκατομμύρια. Οι περισσότεροι συνάδελφοι, όπως και εγώ φαντάζομαι, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς θα καταλήξουμε εκεί, από πού θα προέλθουν τα χρήματα και πώς θα τα διαχειριστούμε κυρίως. Εδώ υπάρχει ασάφεια. Γιατί ποιος θα έχει την εποπτεία, ποιος θα ελέγχει το πώς υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά. είναι οι επικρίσεις μας. Παρόλο που βλέπουμε με συμπάθεια την ιδέα αυτή. Έπειτα πρόκειται για πολλά χρήματα. Εμείς θέλουμε να καινοτομήσουμε, θέλουμε να επενδύσουμε. Με, για τις επενδύσεις θα πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Στην Ευρώπη όμως μιλάμε πολύ και για μεταρρυθμίσεις, για έλλειψη κονδυλίων. Εμείς η Ολλανδική Αντιπροσωπεία βλέπουμε θετικά τις επενδύσεις, δείχνουμε συμπάθεια για το επενδυτικό ταμείο, αλλά θέλουμε και εποπτεία και έλεγχο για τη διαχείριση από την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξακολουθήσει, αυτή την εποπτεία δηλαδή να την έχει η Ευρώπη για την υλοποίηση των επενδύσεων. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος Χέλμουτ Μαρκόφ, Γερμανία. Ο κύριος Κίμον Σαντσί, παρακαλώ, από τη Φιλανδία να ετοιμάζεται. Κύριε Χέλμουτ Μαρκόφ. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε η επένδυση των δημοσίων προϋπολογισμών ε, έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητος λόγων. Τώρα θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να δίνει εγγύσεις για να ε, προκαλέσει ιδιωτικές επενδύσεις. Μία επιχείρηση δεν νομίζετε ότι θα περιμένει να αποκομίσει και όφελος. Τουλάχιστον τόσο όσο και τώρα. Δηλαδή, έργα με τα οποία μπορεί κανείς να κερδίσει χρήμα, πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που θα έκανε το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά με κέρδος. Και μετά μας λέτε ότι έχετε έξι ανεξάρτητους σοφούς σε μια επιτροπή σοφών που θα μελετήσει. Δηλαδή, ανεξάρτητα, ε, μάλλον συμπεριλαμβανομένων των ε, οικονομικών αξιών και αρχών θα δοθούν κάποιες καθοδηγήσεις. Τα κράτη-μέλη με την καλύτερη κατάσταση στα δημοσιονομικά τους θα έχουν ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις από ότι εκείνα όπου το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό. Τρίτη ερώτηση. Γιατί κράτος μέλος να αποφασίσει, να σκεφτεί και να αποφασίσει να δώσει πιο πολύ χρήμα σε αυτό το ταμείο όταν δεν έχει το δικαίωμα να συνδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει τη διαχείριση του χρήματος αυτού, γιατί θα είναι άλλα τα οικονομικά κριτήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και Μοσάση από τη Φινλανδία και ο κύριος Γιώργη Άντενσον της ε, Σουηδίας, παρακαλώ να ετοιμάζετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι χρειάζονται όντως επενδύσεις στην Ευρώπη. Όμως πρέπει οι, ευ... επενδύσεις να είναι πάντα παραγωγικές. Άρα χρειάζεται και ζήτηση από την αγορά στην Ευρώπη και ανταγωνιστικότητα για μας στο παγκόσμιο σκηνικό. Πρέπει να δούμε επίσης αν χρειάζονται επιπλέον μέσα. Ή αν αρκεί το, ευρωπαϊκό σχέδιο, το σχέδιο Juncker, εγώ αμφιβάλλω. 0,5% επιτόκιο έχει για το δανεισμό της Φινλανδία, άρα πρόβλημα δεν έχει η ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαθέτει αρκετή ρευστότητα στην αγορά, άρα τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν και να αρκούν. Όταν λέμε κάθε μέσον για να βελτιωθούν οι επενδύσεις και η απασχόληση, εγώ κάπως ανησυχώ γιατί φτιάχνουμε φούσκα. Φούσκα η οποία μπορεί να σκάσει απότομα και να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Θέλω επίσης να επενθυμίσω ότι έχουμε συγκρουόμενους στόχους στην Ευρώπη. Μικρές επιχειρήσεις, επί παραδείγματι. Η διαθεσιμότητα των δανείων είναι θετική αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα όμως είναι οι τιμές. Γιατί είναι υψηλέ τιμέ για τι μικρότερε επιχειρήσει, Μα γιατί το ορίζουν αυτό, το προκαλούν αυτό οι ρυθμίσει που έχουμε, η νομοθεσία η τραπεζική που έχουμε. Δηλαδή, από τη μια αυξάνουμε τι τιμέ, και εμποδίζουμε τις επενδύσει και από την άλλη προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις ενισχύσεις, τι επενδύσει. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν πρόκειται να αναλάβουν κίνδυνο για τις ε, επιχειρήσεις αυτές. Το κίνδυνο πρέπει να αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη. θα πρέπει να είναι το 60% το δημόσιο χρέος και αυτό πρέπει να είναι απαράβατος κανόνας. Το πακέτο είναι καλό όπως έχει, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι χρειάζεται εμπιστοσύνη στην οικονομία. Πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις πανικού και αυτό αφορά και την ελληνική περίπτωση, στα χέρια μας είναι. Η προβλεψιμότητα της νομοθεσίας είναι πολύ σημαντική, όπως και όσο το δυνατόν πιο ισχνές ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ, Σάνση. Σόν, Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Παλά, παρά μια νυχτή νομισματική πολιτική, έχουμε πολύ χαμηλό επίπεδο επενδύσεων και ίσως γι' αυτό η πρωτοβουλία της Επιτροπής θεωρείται τόσο ευπρόσδεκτη. Έχει συμβολικό χαρακτήρα πάνω απ' όλα στην τρέχουσα κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και να ξαναξυπνήσουμε εμπιστοσύνη για το μέλλον, για τον πολίτη. Πολλοί μίλησαν ε, για τις θετικές επενδύσεις, το πνεύμα, το ρόλο των επενδυτών για να ανακινήσουν επενδύσεις και ανάπτυξη. Πολλοί μίλησαν για τη σημασία της ε, αποδιάρθρωσης της, ε, των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα όπου έχουμε και τη βασική πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της ιστορικής αγοράς. Ο λανθάνων αλλά και διαρκώς ενισχυόμενος προστατευτισμός είναι ο κίνδυνος εδώ. Πρέπει να προχωρήσουμε με περισσότερο άνοιγμα, διαφάνεια, άνοιγμα και στις ξένες επενδύσεις, άνοιγμα προς τον έξω κόσμο, που θα εξασφαλίζει ότι κάθε είδους επένδυση θα μπορεί να φτάνει και να υλοποιείται στην Ευρώπη. Αυτή είναι η έκκλησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή είναι η έκκλησή μου προς τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ουσιώδους ανάγκης ε, να αποτραπεί η ύψωση νέων φραγμάτων, φραγμών από τον προστατευτισμό εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να ανοιχθούμε στις νέες επενδύσεις. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Άντρε ήταν ο τελευταίο στον κατάλογο των ομιλητών μας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους στο πάνελ, αρχικά στον κύριο Μοσχοβίση, ώστε να μπορέσει να απαντήσει και στο μετά στον κύριο Αρτουή για τις τελικές του παρατηρήσεις και για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ο, ο Μοσχοβησή φτάνουμε στην ολοκλήρωση της συζήτησης. Ε, ε, βλέπουμε την προσήλωση και την, ε, το ενδιαφέρον όλων των συναδέλφων Και καταλαβαίνω βέβαια και τις απορίες και τις αμφισβητήσεις και τους προβληματισμούς. Είναι απόλυτα θεμητά όλο αυτό. Αυτό το σχέδιο το θελήσαμε και το συλλάβαμε πολύ γρήγορα. Το πιστεύουμε και ε, το προωθούμε με όλη μας την ε, ενεργητικότητα. Αλλά ε, βέβαια ξέρουμε ότι θα κριθούμε επί των αποτελεσμάτων. Και γι' αυτό και τα ερωτήματα που ετέθησαν εδώ είναι απόλυτα νόμιμα και σκόπιμα. Ε, καταρχήν, για το στόχο των ε, σχεδίων αυτών. Είναι, δεν είναι πρώτη φορά και δεν θα είναι και η τελευταία. Ε, να δούμε ποιες θα είναι οι επενδύσεις που θα μπορούν να γίνουν και για ποια σχέδια. Εμείς θέλουμε να επενδύσουμε ώστε να έχουμε αντίκτυπο στην οικονομία, στις ανεργίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδεια, παιδεία, ε, μεταφορές και σχετικές υποδομές. Ξέρω πως οι ενάγκες των χαρών μελών για όλα αυτά είναι πολλές και διάφορες, ποικίλουν και θα απαντήσουμε στις ανάγκες αυτές, αλλά θα το κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων. Ε, κάτι ακόμα το οποίο συχνά επανήλθε είναι το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα στο σεβασμό των ε, κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητα αλλά και των αναγκών ε, σε επενδύσει. Έχουμε κανόνε που είναι αρκετά πρόσφατοι και μάλιστα και δεν θέλουμε να του αλλάξουμε. Δεν θέλουμε να του αλλάξουμε τώρα γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ε, μια επιτακτική ανάγκη που είναι η εξυγίανση. Αλλά οι κανόνε αυτοί ε, περιέχουν κάποια ευελιξία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό είναι και το νόημα τη ανακοίνωση. Δεν θέλουμε να επανεφεύρουμε κανόνες, δεν θέλουμε να αρνηθούμε το σύμφωνο, ε, στο εσωτερικό του συμφώνου θέλουμε να, κάνουμε, να δώσουμε κάποιες ερμηνείες ώστε να είναι αυτές ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Την ανακοίνωση αυτή σας καλώ να την μελετήσετε γιατί είναι σαφής, μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται τα διάφορα κράτη-μέλη, κατά πόσο δηλαδή είναι στο τμήμα το διορθωτικό ή το προληπτικό. Τώρα, σημασία που δίνουμε στη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ το, από, τότε που εγκρίθηκαν το διπλό και το ξαπλό πακέτο και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων για την εκπόνηση των πολιτικών. Το Ευρωκοινοβούλιο τακτικά ενημερώνεται και διαβουλευόμαστε μαζί του. Πέρα από αυτό όμω βρίσκεται στο επίκεντρο τη νομοθετική διαδικασία. Και επίση στη διάρκεια τη ανάληψη δεσμεύσεων, ε, όταν βρισκόμαστε δηλαδή σε δύσκολη κατάσταση ε, σε οποιαδήποτε χώρα μέλη, έχουμε άμεσα επαφές μέσω του μόνιμου οικονομικού διαλόγου ώστε ε, να μπορούμε και μάλιστα οι επίτροποι ερχόμαστε εδώ για να έχουμε άμεση επαφή. Κάθε επίτροπος όταν έρχεται και επισκέπτεται ένα κρατός θα πρέπει αυτό να το έχει υπόψη και να δώσει λογαριασμό για τα όσα έγιναν εκεί. Χτες έφτασα στην Γερμανία και επισκέφθηκα και τον Bundestag που είχα επαφέ με διάφορου εκπροσώπους πολιτικών ομάδων, όχι τη μία ή την άλλη, όλες τις ομάδες. Και η Κομισιόν είναι, ε, έχει ρητό το να είναι διαθέσιμη για όλου. Τέλο, κάτι ευρύτερο. Το θέμα θέμα της σημερινής μας συζήτησης αφορούσε το Ευρωπαϊκό New Deal. αυτό το σχέδιο το επενδυτικό είναι το Ευρωπαϊκό New Deal. Όχι, δεν ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είμαστε ε, διαυγείς και ε, ρεαλιστές. Πιστεύω ωστόσο πως βρισκόμαστε σε σημείο καμπή. Στις πέντε προηγούμενες ε, χρονιές η Ευρώπη αντιμετώπισε την οικονομική κρίση και το κύριο πρόβλημα ήταν και το γνωρίζετε πολύ καλά και όλοι το ξέρει για τον προκατοχό μου, ε, το πρόγραμμα ήταν να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη, να εγγυηθούμε την ε, οικονομική σταθερότητα και ό,τι και κάναμε. Και εγώ ήμουν υπουργό Οικονομικών. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρήσαμε. Ε, έχουμε μηχανισμούς τώρα, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Τραπεζική Ένωση. Δεν ήταν εύκολο, προσκέφταμε τα προγράμματα από όπου επέρχονται περισσότερες χώρες ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ισχύ του τραπεζικού συστήματο. Τώρα το, η πρόκληση είναι διαφορετική. Αναγνωρίζουμε μια ανάκαμψη, αλλά είναι πολύ αργή και αδύναμη. Δεν αρκεί και δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε με μια οικονομία τόσο αδύναμη, μικρό πληθωρισμό και υπερβολικά πολύ ανεργία, γιατί μετά ο λαϊκισμός αρχίζει και κερδίζει έδαφος και το ξέρουμε η Ευρώπη θα πρέπει να κριθεί και να δείξει τις αρετές της μέσω των αποτελεσμάτων και θέλουμε να δοθεί ένας νέος δυναμισμός στην οικονομία μας και γι' αυτό και θέλουμε ε, πολιτική, δημοσιονομική που να είναι προσαρμοσμένη σε όλα αυτά και έχω μιλήσει γι' αυτό, για την ευελιξία. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν ε, ε, μεταρρυθμίσεις διευθυντικές αλλά και να υπάρξει και ε, η ορθότερη λειτουργία των εσωτερικών αγορών, γιατί δεν είναι μία η εσωτερική αγορά, υπάρχουν ακόμα προβλήματα και φράγμοι ανάμεσα στις εσωτερικές αγορές που έχουμε. Και έπειτα, Είδαμε όλοι οι Ευρωπαίοι πως ο Μάριο Ντράγκη ενήργησε προς το συμφέρον ολόκληρη της Ευρώπης. Μικρός, ισχνός ε, πληθωρισμός και προβλήματα ανάπτυξης. Ε, ε και έπειτα, αυτό το σχέδιο το επενδυτικό είναι μια συμβολή σε αυτή τη νέα προσέγγιση που όντως θα πρέπει να επιτρέψει και θα επιτρέψει με βέβαιος ε, μεγαλύτερη ανάπτυξη. Είμαστε πολύ αποφασισμένοι <coughs> με βέβαια τον απαραίτητο ρεαλισμό και ξέρουμε πως δεν θα κριθεί το σχέδιο επενδύσεων από Γιούνκερ από το σχεδιασμό του, αλλά από τα αποτελέσματά του και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Και γνωρίζουμε όλοι ποιες είναι οι ευθύνες μας. Ένα σχέδιο δεν είναι αποτέλεσμα και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας με βάση τα αποτελέσματα που θα επιτύχουμε. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μοσχοβησή. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αρτουή να απαντήσει, να κάνει σχόλια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είπα πράγματι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ προσεκτικό σε όλες τις παρατηρήσεις, όλα όσα ακούσαμε σήμερα το πρωί. Και ότι φυσικά και θα τα λάβουμε υπόψη μας την προετοιμασία της ψηφοφορίας του νομικού εργαλείου που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εφαρμόσει την ιδέα αυτή του επενδυτικού πακέτου. Θέλω να απαντήσω στον κύριο και ο οποίος με ρώτησε για, τη την διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Θέλω να επανέλθω λίγο στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη, η οποία για μία δεκαετία λειτουργήσε με κάτι σαν κυβέρνηση, σχεδόν κυβέρνηση, που είναι το Eurogroup. Το Eurogroup πράγματι δεν κατάφερε να ελέγξει πλήρως την κατάσταση. Η κατάσταση κατέληξε στην κρίση δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη. Είδαμε σε τι βαθμό τα μέλη της Ευρωζώνης είχαν ειδική ευθύνη που δεν είναι η ίδια με τις υπόλοιπες χώρες μέλη, με τις υπόλοιπες από τα 28. Είδαμε επίσης ότι όταν χρειάστηκε βοήθεια δεν είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, δεν είναι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή που δίνουν διμεριδάνεια. Όχι, είναι οι χώρες της Ευρωζώνης και είναι τα κοινοβούλια της Ευρωζώνης τα οποία ε, γράφουν στους λογαριασμούς τους τις απαραίτητες πιστώσεις για να βοηθήσουν εκείνους που βρίσκονται σε δυσκολία. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον με την Ευρωζώνη. Και αυτό δικαιολογεί γιατί τα κοινοβούλια της Ευρωζώνης πρέπει να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακυβέρνηση. Γιατί, γιατί έχουμε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το κεφάλαιο βρίσκεται στα χέρια των μελών της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πράγματι έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει και μερικές φορές ξεπέρασε και τόσα προβλέπουν οι συνθήκες. Αλλά για να κάνουμε το περίφημο policy mix, το πολιτικό μείγμα εκείνο δημοσιονομικής, οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής όπως κάνουν στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο συνομιλητής μας, είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος της Ευρωζώνης. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί, αυτή δηλαδή η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Κάνουμε μια διάκριση λέτε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από εκείνες που θέλουν να μείνουν εκτός ενιαίου νομίσματος, όλες οι χώρες κάποια στιγμή μπορούν να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Έχουμε και θέμα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο Ευρωπαϊκός Μεχανισμός Σταθερότητας είναι κάτι το οποίο σήμερα δεν ελέγχεται από κανένα κοινοβούλιο. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Θα πρέπει να δώσουμε δημοκρατική νομιμότητα στην ε, κυβέρνηση της Ευρωζώνης. Έτσι ελπίζω να έρθουν όλοι οι φόβοι όσον αφορά την διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να υπάρχει καμία υπόνοια έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Ελπίζω να το καταφέρουμε αυτό. Και αυτή η εμπιστοσύνη θα οδηγήσει και σε εμπιστοσύνη των πολιτών μας στο μέλλον, στην Ευρώπη και στο επενδυτικό σχέδιο Juncker. Σας ευχαριστώ πολύ σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Αρτουή. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω το προνόμιο όσο προεδρεύων να καταλήξω σε μερικά συμπεράσματα. Πρώτον, και οι δύο κύριοι ομιλητέ, αλλά και οι παρατηρήσει των μελών των κοινοβουλίων υπογραμμίζουν τον κατεπήγοντα χαρακτήρα για την υλοποίηση και την ανάγκη για υλοποίηση των μέτρων. Επίσης ότι πρέπει άλλα ε, άλλες ε, οικονομίες που βρίσκονται μπροστά ή ε, αναπτύσσονται ταχύτερα, πρέπει και εμείς αντίστοιχα να προχωρήσουμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το New Deal για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμηλό επίπεδο επενδύσεων. Αυτή είναι τόσο η αιτία όσο και το αποτέλεσμα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκής οικονομίας και της χαμηλής ελκυστικότητας της τάσης της ως προορισμού για επενδύσεις. Φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο και ρυθμιστικά περίπλοκο το περιβάλλον για τις επενδύσεις στην Ευρώπη και έτσι αυτές σπέβδουν σε άλλες αγορές όπως οι ασιατικές ή η Βραζιλία. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε το στόχο, να γίνουμε πιο ελκυστικοί για τις ε, επενδύσεις, να δώσουμε μια θετική εικόνα πρόσβασης, μια θετική πρόσβαση για τις επιχειρήσεις, για το, η παραγωγή του κέρδους, για την εξασφάλιση μιας μεγάλης αγοράς με την κατάργηση των φραγμών μεταξύ των οικονομιών μας. Η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει έναν ανταγωνισμό, αλλά όχι προς τα κάτω, όχι περικόπτοντας. Βεβαίως θα πρέπει να ανταγωνιστούμε, αλλά με όρους την ποιότητα και την υψηλή προσθεμένη αξία δεν χρειαζόμαστε απλώς και μόνο θέσει εργασίας. Χρειαζόμαστε υψηλής ποιότητας και με πολύ καλές αμοιβέ θέσεις εργασίας. Όπως είπε και ο Επίτροπος Μοσκοβισή, οφείλουμε να επενδύσουμε ευθυγραμμισμένοι με τις ε, ανάγκες του μέλλοντος, με την καινοτομία, με την ανάπτυξη, με τις υποδομές. Είπε και ο κ. Σαντέρα ότι θα πρέπει να δούμε τις επενδύσεις ως ε, ένα βήμα για το μέλλον και όχι ως απλά έξοδα. Για τις επικρίσεις, ότι μπορεί να μην είναι παρκές αυτό το σχέδιο ή ότι θα πρέπει να είναι πιο οικολογικό ή πιο αυστηρό στην, στον προσδορισμό των όρων. Βεβαίως όλα μπορούν να βελτιώνονται, τα πάντα μπορούν να βελτιωθούν. Αλλά πρέπει να έχουμε την ευκαιρία για το μέλλον, να έχουμε μια Ευρώπη πιο καλή, πιο αποτελεσματική πιο λειτουργική και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε ενθάρρυνση και στην καινοτομία και στην αποτελεσματική δράση που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη. Καλό θα ήταν να συζητούμε ακόμα για μερικά χρόνια. Καλό θα ήταν να, να κοιτάξουμε τον ιδεώδη, το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αλλά νομίζω ότι το άριστον θα ήταν να αρχίσουμε να καλύπτουμε το χαμένο έδαφος στο παγκόσμιο ανταγωνισμό και να συνεργαζόμαστε κατά τρόπο αποτελεσματικό και καλό μεταξύ μα εκεί που θεωρούμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύση προς την ορθή κατεύθυνση. Τέλος. τα κράτη-μέλη πρέπει και να συμμετάσχουν και να υιοθετήσουν αυτά τα έργα. Δεν μπορούν οι επενδυτές να έχουν να κάνουν μόνο με Βρυξέλλες και Στρασβούργα. Κολίγκα είναι αυτή, η Αβινιό είναι αυτή, το Παρίσι είναι αυτό, η Νάπολη είναι αυτή. Κάθε μικρή πόλη, κάθε όχι τόσο μεγάλη πόλη της Ευρώπης πρέπει να συμμετάσχει. Και να ξέρουν οι επενδυτές ότι στα έργα αυτά στέκονται παραστάτε στα κράτη-μέλη. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την ισχυρή μας συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων, άσχετα αν δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ, συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού. Διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στην προσοχή μα συνεδρία στι 2 το μεσημέρι για την παρούσα σύνοδο συνεδρία. σα ευχαριστώ πολύ όλου και όλε. τους ομιλητές μας από το Προεδρείο, τους συναδέλφους που μοιράστηκαν μαζί μας στις θέσεις τους, αλλά και εκείνους που απλώς άκουσαν και φαντάζομαι συνέλεξαν νέες και καινούριες και καλές ιδέες. Εν τέλει. Με χαρά. Κυρίσω, κυρίσοντας το πέρας της ε, συνεδρίας, σας καλώ, ίσως το πιο ευχάριστο κομμάτι σε ένα ε, γεύμα με σάντουιτς, ένα πρόχειρο γεύμα στην, ε, στο χώρο Γεχουντι Μενουχίν, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου στο οποίο βρισκόμαστε και μετά θα τα ξαναπούμε στις 2. Προς το παρόν σταματάμε.